Συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε. Ξεκινάει η επίσημη συνεδρίαση της Επιτροπής μας, ξαναρχίζουμε. Είναι μεγάλη χαρά μου που σας συναντώ όλους μετά από διακοπές εξαίρετες από ό,τι κρίνω τουλάχιστον από το μαυρισμένο σας στεύμα και το χαμόγελό σας το αποφασιστικό. Νομίζω ότι η χρονιά που θα ζήσουμε θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα για τον προϋπολογισμό, την προετοιμασία του 17 του προϋπολογισμού, όπως επίσης και την ενδιάμεση αναθεώρηση. Και περιμένουμε να δούμε Επίσης και τις προτάσεις για τον προϋπολογισμό της ζώνης ευρώ. Είναι κάτι που το συζητάμε από χθε το απόγευμα. Σας χαιρετώ λοιπόν με πολύ μεγάλη χαρά. Έχετε την ημερήσια διάταξη, το σχέδιο της ημερήσιας διάταξης. Καταρχάς το 6 και το 16 ε, αναβάλλονται. το 11 και το 12 αντιστρέφονται θα εξετάσουμε το 12 πριν από το 11, όπως επίσης και το 14 πριν από το 13. Και τέλος, στο σημείο 20 για τις μεταφορές στον προϋπολογισμό του 16. Ε, θα ασχοληθούμε και με τα θέματα της ασφάλειας. Θα συζητηθεί και κλεισμένο των θυρών τελευταίο Λοιπόν, αν δεν έχετε αντιρρήσεις, <clears throat> θεωρώ ότι η μερίσια διάταξη είναι πλέον δεκτή. Δεν έχω κάποια ανακοίνωση να σας κάνω. Να σας πω ότι μετά από αίτημα του κυρίου Σούλτς, εγώ μετέβη στην Παλαιστίνη στις 18 μέχρι τις 21 Ιουλίου στη Γάζα <clears throat> κανένα μέλος ε, του Κοινοβουλίου δεν είχε πάει εδώ και πέντε χρόνια και πήγα και στην Υπεριορδανία. Αναφέρθηκα για την έκθεση αυτή, βρίσκεται στην ιστοσελίδα μου η αναφορά. Δεν πήγα ως πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών, αλλά ο πρόεδρος Σούλτς θέλησε με την ιδιότητά μου αυτή να επισκεφθώ την Παλαιστίνη. Έχετε τα πρακτικά των συνεδριάσεών μας της 15ης και τις 30ης Ιουνίου, όπως και τις 4ης, 11ης και 12ης Ιουλίου. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, τα πρακτικά αυτά θεωρούνται δεκτά. Εάν ο Γενικός Εισηγητής του 17 είναι έτοιμος, θα του δώσω το λόγο. Θα πάρει το λόγο και ο κύριος Τάραντ για τα υπόλοιπα τμήματα. Κύριε Γκάιερ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την εισαγωγή αυτή και να συμφωνήσω και εγώ μαζί σας, να ευχηθώ και εγώ στους συναδέλφους ε, ε, καλό φθινόπωρο, ελπίζω να περάσετε καλά το καλοκαίρι και να ξεκουραστήκατε καλά γιατί θα το χρειαστείτε. Το δεύτερο ήμιση του έτους βλέπετε σε ό,τι αφορά θέματα προπολογισμού θα μα φέρει αντιμέτωπους με διάφορε ιδιαίτερε προκλήσει. Δεν ξέρω κατά πόσο ο προπολογισμό το 2017 ε, είναι ένα από τα θέματα αυτά. Γιατί το Συμβούλιο το οποίο αναγκάστηκε να καταλήξει σε μια τοποθέτηση υποχρονική πίεση κάνει λίγο πράγματα όπω τα είχαμε συνηθίσει, αλλά έχει αλλάξει και κάποιε πρακτικέ στο παρελθόν. κοιτώντα λοιπόν το τι έχει αλλάξει, ως προς τη συμπεριφορά του Συμβουλίου. Διαπιστώνουμε και αξίζει τον κόπο να το σημειώσουμε αυτό ότι οι αλλαγές που προτείνει το Συμβούλιο στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε έχουν ε, αποτύχει. Υπάρχει λοιπόν διαφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Επιτροπής σε ό,τι αφορά ε, ζητήματα που αφορούν το 1% του προϋπολογισμού στις πληρωμές. Δηλαδή ουσιαστικά τσακωνόμαστε για 1,3 δις ευρώ για τέτοιους όγκους, για τέτοιες ποσότητες. Ε. Άρα τι εξυπηρετεί αυτό, αναρωτιέται κανείς. Και εγώ αναρωτήθηκα ειλικρινά όταν έλαβα την πρόταση του Συμβουλίου, την οποία και δημοσίευσε το Συμβούλιο λίγο πριν τις θερινές διακοπές και σε μια πρώτη ανακοίνωση τύπου αυτό που δήλωσα είναι κατηγόρησα μάλλον το Συμβούλιο για αυτά που κάνει, γιατί ουσιαστικά αποδυναμώνει τα εργαλεία αντιμετώπιση κρίσεων, τα οποία το ίδιο το Συμβούλιο είχε ορίσει ως στοιχεία προτεραιότητας. Αν θέλουμε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να φροντίζει τα μεγάλα ζητήματα και αν θέλουμε να συμφωνήσουν όλα τα θεσμικά όργανα διότι ο στόχος θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη και η απασχόληση. Έμα τότε θα πρέπει τα εργαλεία τα οποία διαθέτει προς την διαθέτει προς την κατεύθυνση αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστούν όντως πολιτική προτεραιότητα και αυτά να αποτελούν το επίκεντρο της πολιτικής μας. Και στην κατηγορία λοιπόν 1α για να δούμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για περικοπές. Όλοι συμφωνούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση άλλωστε ότι η επίλυση του μεταναστευτικού, το είναι ένα θέμα που μας ε, απασχολεί ιδιαιτέρως εδώ και δύο χρόνια, είναι σημείο προτεραιότητας. Και το Συμβούλιο δεν κάνει περικοπές στην κατηγορία 3. Αυτό είναι λογικό, γιατί από αυτό ωφελούνται πιο πολύ τα κρατημέλη, σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, γιατί εδώ περιλαμβάνονται όλα τα εργαλεία τα οποία ε, συμβάλλουν στην ιστορική πολιτική, αλλά κάνει περικοπές που στην κατηγορία 4, σε ό,τι αφορά την εξωτερική αποδυνητική που άπτεται της αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Όλα λοιπόν αυτά τα εργαλεία της πολιτικής γειτονίας, σε ό,τι αφορά και την Τουρκία, σε ό,τι αφορά την προενταξιακή βοήθεια, με αυτά προσπαθεί κάπω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα αντιμετωπίσει κάπως πιο ευρέως. Κάναμε λοιπόν μια εκτεταμένη έρευνα σε ό,τι αφορά και τη δεύτερη δόση της ε, βοήθειας που έχουμε υποσχεθεί προς την Τουρκία για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Αυτή είναι η τοποθέτησή μου και θεωρώ ότι από πολιτική άποψη έχει σοβαρά επιχειρήματα που την υποστηρίζουν. Νομίζω λοιπόν ότι οι συνάδελφοι από την Επιτροπή ανάπτυξη, από την ε, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, θα τα πούνε αυτά και πολύ πιο έξω από τα δόντια. Άρα ουσιαστικά για ένα μικρό σχετικά ποσό τσακωνόμαστε. Και όταν συνομιλούμε με τους εκπροσώπους του Συμβουλίου και τοποθετούνται κάπως, μας ε, αναφέρουν ποιες ήταν λίγο πολύ οι τοποθετήσεις μεταξύ των κρατών μελών στο Συμβούλιο. Αυτό ασφαλώς δεν μας προκαλεί έκπληξη και δεν είναι και κάτι καινούριο άλλωστε, ότι οι καθαροί εισφορείς, τα κράτη που είναι καθαροί εισφορείς, επιμένουν στα συγκεκριμένα περιθώρια, όσο περιορισμένα κι αν είναι, ενώ οι χώρες οι οποίες ουσιαστικά λαμβάνουν χρήματα έχουν ε, ιδιαίτερο συμφέρον σε ό,τι αφορά τα περιθώρια αυτά. Το θέμα όμως, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι τα περιθώρια εδώ. Πρόκειται για μια κρίση την οποία ε, δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε ενδεχομένω, αλλά μια κρίση για την οποία θέλουμε να δαπανίσουμε ένα δις ευρώ. Τι κρίση είναι αυτή λοιπόν σε τελική ανάλυση θα πρέπει ο, οι καθαροί εισφορείς ε, να προβούν σε μεγαλύτερη αποταμίευση, σε περικοπές πιο μεγάλες από αυτές που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και όταν μιλάμε για τέτοιες ε, περικοπές, ε, μιλάμε για το εθνικό επίπεδο. Ακόμα και το ίδιο το επιχείρημα του Συμβουλίου ότι αν κάνουμε κάποιες περικοπές θα δημιουργηθούν περιθώρια και παθηματικά για άλλε άλλες καταστάσεις ενδεχόμενης ανάγκης και αυτό μπάζει. Θα ήθελα να είμαστε ειλικρινείς λοιπόν στην επιχειρηματολογία μας γιατί δεν απορρίπτουν το σχέδιο προϋπολογισμού από το Συμβουλίο. Ο προπολογισμό είναι πιο υψηλός από το 2016. Αυτό που κάνουν είναι ότι δεν ακολουθούν 100% τις αυξήσεις που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με μία και μοναδική εξαίρεση, αν δεν κάνω λάθος, στην κατηγορία 4 για την εξωτερική πολιτική. όπου το ποσό που προτείνει το Συμβούλιο είναι κάτω του 2016. Αυτό πραγματικά είναι ανήκουστο. Έχουμε πολιτικές προτεραιότητες, τις οποίες και υλοποιούμε. Ουσιαστικά αυτό λοιπόν είναι αντίθετο με την ίδια την επιχειρηματολογία του ίδιου του Συμβουλίου. Δεν γίνεται και το, την ολόκληρη και το σκυλοχορτάτο. Δεν μπορούμε και να θέλουμε να υλοποιήσουμε πολιτικές αρχές και να προσπαθούμε ε, παράλληλα κάποια κράτη-μέλη να ξοδέψουν και λιγότερα. Πώς θα γίνει αυτό. Έτσι λοιπόν έχει διαμορφωθεί το έγγραφο εργασία, το οποίο και προετοίμασα την προηγούμενη εβδομάδα και σας διαβίβασα άλλωστε σε ό,τι αφορά την ανάλυση της τοποθέτησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τώρα, το ποια θα είναι τα πολιτικά συμπεράσματα, τα πολιτικά απορίσματα τα οποία θα πρέπει να εξαγάγουμε από την θέση του Συμβουλίου, δεν θα σας εκπλήξει το γεγονός ότι σε μεγάλο βαθμό σας προτείνω, και αυτό συνάντηκε και με την παράδοση των προκατόχων μου και των ε, συναδέλφων που προηγήθηκαν ως εισηγητές ε, για τον προϋπολογισμό, σας προτείνω λοιπόν στο 1α, στην κατηγορία 1α να αξιοποιήσουμε όλο το περιθώριο για την ε, χρηματοδότηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Και σας προτείνω λοιπόν να χρησιμοποιηθούν τα περιθώρια έκτακτης ανάγκης, τα contingency margins. για την αντιστάθμιση που συμφώνησαν το Συμβούλιο και η Επιτροπή για την χρηματοδότηση του Ταμείου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Υπάρχει ένα σημείο στο οποίο ενδεχομένω δεν είμαι βέβαιο, αλλά θα σα το αναφέρω. Είτε θα το συζητήσουμε και θα το αποφασίσουμε μεταξύ μα, είτε θα τσακωθούμε. Είναι φλεγόμενο το ζήτημα αυτό. Υπάρχει λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, μια κοινή πιλωτική δράση η οποία προτείνεται αλλά και από το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υποστηριχθεί. Αλλά κοιτάξτε, βασικά πρόκειται για μια πρόταση γερμανογαλλική. Μια πλειοτική λοιπόν δράση να ξεκινήσει στα πλαίσια του τρέχοντος αυτού προϋπολογισμού για την αξιοποίηση της συνεργασίας ε, της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Εξοπλισμών. που θα προαπαιτούσε περίπου 90 εκατομμύρια. Αυτό υπολογίζεται στην παρούσα φάση και αυτό θα εντασσόταν ε, στον τίτλο 1α. Αυτή η πιλωτική δράση, κοίτοντας λοιπόν τον όγκο των πόρων που θα χρειαζόταν, έχω να πω ότι αναρωτιέμαι τρία πράγματα. Τρεις ερωτήσεις πρέπει να θέσουμε. Πρώτη ερώτηση. που μπορεί να συζητηθεί σε όλε τι επιτροπέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο Συμβουλίο κατά πόσον η ενίσχυση μιας πρωτοβουλίας ε, στα πλαίσια της ΚΕΠΑ μέσω της βιομηχανίας εξοπλισμού είναι αυτό που πραγματικά χρειάζεται η Ευρώπη φέτος. Αυτό μπορεί κανείς να το συζητήσει. Η πολιτική μου λοιπόν άποψη και το πολιτικό μου ένστικτο είναι ότι μάλλον όχι. Δεν είναι αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη φέτος. Αλλά φυσικά έχω διάθεση συμβιβασμού. Μια πιο, άλλη, μια πιο σοβαρή ερώτηση είναι η εξή. Αν τυχόν καταλήξουμε σε πολιτική συμφωνία για το γεγονός ότι η πολιτική ασφάλειας και η εξωτερική πολιτική θα πρέπει να αποτελέσει το μοχλό που θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να περάσει το επόμενο επίπεδο της αντιμετώπισης της ευρωπαϊκής κρίσης και αν καταλήξουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι αυτό είναι κάτι το ευκταίο ω υπεύθυνη χάραξη του προπολογισμού, θα πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε πώ θα χρηματοδοτηθεί αυτή η δράση. Εδώ λοιπόν δεν θα σας προκαλέσει έκπληξη το γεγονός ότι ως τώρα δεν έχω ακούσει ιδιαίτερα σωστές προτάσεις και δεν είμαι δεθυμένος να ακολουθήσω καμία από τις προτάσεις που έχω ακούσει. Συμφωνούμε ότι ο προπολογισμό ήδη σήμερα δεν είναι σε θέση να υλοποιήσει τους πολιτικούς στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα ικανοποιητικό βαθμό. Και στην κατάσταση λοιπόν αυτή όσο έχει αγαπητοί συνάδελφοι, έρχεται ένας νέος πολιτικός στόχος, μία νέα πολιτική πρωτοβουλία, επιπρόσθετα εγώ στο Κοινοβούλιο συμμετέχω από το 2009 και μετά, αλλά η πρώτη ερώτηση που έχω να σας θέσω είναι θυμάται κανείς από εσάς ποτέ μια πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για μια επιπρόσθετη ε, ανάθεση καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνοδεύτηκε ποτέ με αύξηση της χρηματοδότησης. Εγώ δεν το θυμάμαι ποτέ. Και γι' αυτό λοιπόν στις ανεπίσημες συναντήσεις που είχα είπα ναι, Κάντε τα όλα αυτά. Δεν λέμε. Αλλά υπάρχει για την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας ένα εργαλείο μεταξύ των κρατών μελών το οποίο λειτουργεί σωστά. Και δεν είμαι δεθειμένος να χρησιμοποιήσω να... Το, τη χρηματοδότηση αυτή για μια πολιτική δράση η οποία τώρα θα ξεκινήσει. Τώρα ξεκινάει, το τονίζω αυτό. Θα συνεπάγεται πολύ περισσότερες πολιτικές ε, δράσεις. Εγώ δεν είμαι διτεθειμένος να επιβαρύνω με μια επιπρόσθετη πολιτική πρωτοβουλία ένα ήδη επιβαρημένο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Αν μιλάμε για ποσά, αυτό θεωρώ ότι υπερέχει ως επιχείρημα. Θα πρέπει δηλαδή να σφαγιάσουμε πολλά από τα project τα οποία υπάγονται στον τίτλο 1 για να δώσουμε σώμα και σάρκα και οστά στην πρωτοβουλία αυτή. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Θέλουμε όμως να το κάνουμε αυτό. Γιατί αυτό θα ανοίξει το δρόμο και για άλλε τέτοιε παρόμοιε πρωτοβουλίε. Και βρισκόμαστε στα πλαίσια μια συζήτηση όπου θα μπορούσαμε και για τη μεσοπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμο το μεσολυμικό πλαίσιο να πούμε ότι εντάξει αγαπητά κρατημέλη, αν θέλετε να συνεργαστούμε προ την κατεύθυνση αυτή. <clears throat> Και όντω ε, θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε την ε, βιομηχανία εξοπλισμών υπάρχουν τα σωστά επιχειρήματα. Δεν συμφωνώ απόλυτα, αλλά εν περιπτώσει τα κατανοώ. Αν λοιπόν στο σημείο αυτό δεν επιτύξουμε την απαραίτητη προσοχή και δεν ε, πάρουμε σοβαρά τις ε, πρωτοβουλίες στα πλαίσια της ΚΕΠΑ, αν δεν πούμε στο Συμβούλιο ότι κοιτάξτε εδώ έχουμε επί της αρχής, όχι επί του υπηρχομένο επί της αρχής έχουμε αντιρρήσεις. Και θέλουμε να το συζητήσουμε αυτό επισταμένως μαζί σας για το πώς θα α, υλοποιούνται όλα αυτά και μελλοντικά. Προτού περάσουμε στα θέματα περιεχομένου, ε, θεωρώ ότι ανοίγουμε ένα παραθυράκι αγαπητοί συνάδελφοι, το οποίο δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ξανακλείσουμε. Ποτέ δεν θα μπορέσουμε να το ξανακλείσουμε, το ξαναλέω και δεν θα καταφέρουμε καν να χρηματοδοτήσουμε την πρωτοβουλία αυτή. Για αυτό λοιπόν προτείνω αυτή την πρωτοβουλία να δούμε πώς ε, θέλει να αξιοποιήσει το Συμβούλιο τα χρήματα οικονομικά αυτά μέσα. Και αν πιστεύετε μπορεί να βρει, εντάξει. Για το 1β τώρα. Κατανοώ ότι πολλοί από εσά ε, έμειναν έκπληκτοι, δυσάρεστα έκπληκτοι, δυσάρεστη έκπληξη, όταν είδαν τα αριθμητικά στοιχεία, τα ποσά που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί σε σχέση με τον προπολογισμό του 2016, ουσιαστικά ήταν ε, μια μείωση 1 τέταρτο, κατά 1 τέταρτο σε σχέση με τα, τον προπολογισμό του 2016. Αλλά θα πρέπει να αναλύσουμε τα ποσά αυτά και θα πρέπει κατά την ανάλυση αυτή να έχουμε ένα πράγμα υπόψη, ότι η ευθύνη ε, δεν είναι στις Βρυξέλλες. Αυτό δεν προέρχεται από τι Βρυξέλλες. Πολλά κράτη-μέλη σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν καταφέρει να ε, καταθέσουν λειτουργικά προγράμματα προς την ε, Βρυξέλλες, τα οποία να θεωρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μπορούν να ξεκινήσουν. Μα αν δεν υπάρχει τέτοια κατάθεση προγραμμάτων, δεν έχει νόημα να δίνονται οι πόροι αυτοί. Δεν αφαιρούνται πόροι από κανέναν. Υπάρχουν εθνικοί φάκελοι οι οποίοι προβλέπονται για το μεσοπρόθεσμο ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Αλλά θα πρέπει να ακολουθούν προτάσεις λειτουργικών προγραμμάτων που θα ακολουθούν τις πολιτικές ε, συμφωνίες, τους κανόνες που έχουν ε, αποφασιστεί εδώ. Γι' αυτό πιστεύω και παρακαλώ όσοι έχουν πρόβλημα σε ό,τι αφορά τα ποσά αυτά, να κάτσουν να συζητήσουν επισταμένως αυτά με τις ε, κυβερνήσεις και με τις ε, εκάστοτε χώρες για το πώς γίνονται προτάσεις για τέτοια προγράμματα και πώς εγκρίνονται οι προτάσεις αυτές, γιατί εγώ γνωρίζω από συζητήσει με υψηλό βαθμό στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γνωρίζω ότι υπάρχουν ιδιαίτερε ανησυχίε για το γεγονό ότι υπάρχουν πολλά προγράμματα τα οποία δεν μπορούν να εγκριθούν και η πολιτική φαντασία σας φαντάζομαι φτάνει στο το τι θα συμβεί στην επόμενη δημοσιονομική περίοδο σε ό,τι αφορά το επόμενο μεσοπρόθεσμο μεσονομικό πλαίσιο από το 2020 και μετά, τι συζητήσει θα διεξαχθούν μεταξύ Βρυξελών και κρατών μελών, αν η κατάσταση δεν αλλάξει στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, κράτη-μέλη δεν είναι σε θέση να καταθέσουν προτάσεις που να έχουν δυνατότητα να εγκριθούν σε θέματα περιφερειακής πολιτικής. Αυτό μπορεί να σημάνει και το τέλο της περιφερειακή πολιτική, όπω τη γνωρίζουμε σήμερα. Και το λέω ξεκάθαρα ότι αυτό δεν θέλω να συμβεί. Δεν θέλω. Αλλά το θέμα λοιπόν δεν θα είναι να πειράξουμε τα ποσά και τις, ε, τους πόρους γιατί εγώ δεν μπορώ να πω ότι θα πρέπει να δώσουμε πιο πολλά χρήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρχεται και μας λέει ότι δεν ξέρουμε αν καν θα χρειάζονται οι πόροι αυτοί από το 2017 και μετά, γιατί δεν ξέρουμε πολύ απλά αν θα υπάρχει σωστή απορρόφηση από πλευρά. δηλαδή πολιτικής ε, χάραξης του προπολογισμού. Δεν ξέρω κατά πόσον έχει νόημα. Επί το περιεχομένου ανησυχώ ιδιαίτερα για την περιφερειακή πολιτική, αλλά οι ανησυχίες αυτές θα πρέπει να συζητηθούν κάπου αλλού, σε άλλα πλαίσια, όχι στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων αυτών, γιατί αυτό θα έχει και συμβολική αξία, ε, δύσκολη συμβολική αξία. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι είναι αβάσιμες αυτές οι προτάσεις για διαγραφή τέτοιων ποσών όπως προτείνει το Συμβούλιο. Έχει καταθέσει προτάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν οι προτάσει αυτέ. Γι' αυτό λοιπόν εδώ πιστεύω ότι θα πρέπει να επανέλθουμε στα πλαίσια του σχεδίου προεπιλογισμού. και στο 1β εντάσσεται και η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. να ε, ρωτήσουμε και τον κύριο Πρέντα κατά πόσο υπάρχουν συγκεκριμένε ημερομηνίε καταληκτικέ, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μα καταθέσει μια αξιολόγηση τη ε, δράση τη ε, Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων και τα αποτελέσματα που έχει πετύχει ω τώρα. Όσο έχουν οι δομέ σήμερα και όπω εφαρμόζεται η πρωτοβουλία, θεωρώ για παράδειγμα ότι στην Ιταλία τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Αυτό λοιπόν τι θα σήμαινε ότι η πολιτική επιχειρηματολογία που ακούσαμε πέρσι όταν ήταν ο κ. η εισηγητής ήταν πραγματικά εύστοχη. Είπαμε λοιπόν τότε, ας δούμε πώς θα εξελιχθεί η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Έχουμε λοιπόν σχετικά σχετικές ενθαρρυντικές, ε, σχετικά ενθαρρυντικές απαντήσεις στα ζητήματα αυτά που συζητήθηκαν πέρσι φέτος. Ίσως θα μπορούσε να μας πει και ο συνάδελφος τι θα έπρεπε να περιμένουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Αλλά εγώ έχω να πω το εξή. Αν η αξιολόγηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι θετική, θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να αποτυπωθεί και στη διαμόρφωση του προπολογισμού. Και αν πραγματικά το Συμβούλιο πιστεύει στους στόχους για την απασχόληση και την ανάπτυξη που έχει θέσει, δεν θα μπορέσει να πει και όχι. Στον τίτλο 2 τώρα. Να επανέλθουμε σε ό,τι αφορά το σχέδιο του προπολογισμού. Αυτό θα έλεγα. Αυτό θα πρότεινα. Και συμφωνώ να μπορέσουμε να συνεχίσουμε στην, ε, στο Εδώ θα μπορούσε ενδεχομένω να μα μιλήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μα δώσει πιο πολλέ λεπτομέρειε από αυτέ που έχουμε ω τώρα. Τώρα, στον τίτλο 3, το ανέφερα αυτό και στην αρχή. Αυτό, εδώ τα πράγματα, εδώ το Συμβούλιο δεν έκανε μεγάλε αλλαγέ. Αλλά εδώ τα περιθώρια πραγματικά είναι τόσο περιορισμένα Μιλάμε για περικοπές ε, στα προγράμματα από τα πολιτισμικά, στο Creative Euro, στα προγράμματα ανταλλαγών. Όλα αυτά πραγματικά πρέπει να σας πω ότι μου αφήνουν μια πικρή γεύση. Κοιτώντα και τις ε, προτεραιότητες που έχει θέσει, όπως σας είπα, και το Συμβούλιο. Τώρα, στον τομέα 4. Εδώ προτείνω λοιπόν να επανέλθουμε στο σχέδιο προϋπολογισμού και να χρησιμοποιήσουμε το περιθώριο και ανάγκης. Μπορούμε να συζητήσουμε το πού ακριβώς θα γίνει αυτό, αλλά να χρησιμοποιηθούν αυτά τα περιθώρια για την αντιμετώπιση των αιτιών της μετανάστευσης. Από πλευρά αναπτυξιακή πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε όλα σύξυλα. Ούτε να κάνουμε τόσο μεγάλες περικοπές. Θεωρώ λοιπόν ότι οι περικοπές αυτές ενδεχομένω να προκαλέσουν και να οξύνουν κρίσεις. Οπότε δεν έχει νόημα να προσπαθούμε να επιλύσουμε ένα πρόβλημα δημιουργώντας ένα άλλο. Σε ό,τι αφορά την Τουρκία. Σε ό,τι αφορά τις πληρωμές και θα κλείσω μετά θα σας πρότεινα να ε, επανέλθουμε στην πρόταση προπολογισμού και στην ε, κατηγορία 4 να αυξήσουμε τις πληρωμές προκειμένου να ισοσταθμιστούν οι δεσμεύσει και οι πληρωμές. Αυτή λοιπόν η σύντομη ή ίσως και λιγότερο σύντομη κοιτώντα και το ρολόι ανάλυση μου για αυτά που μας κατέθεσε ως πρόταση το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού του 2017 και με χαρά θα ακούσω και τις δικές σας προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γενική Εισηγητά. Μπορεί να ξεκινήσει η συζήτηση. Κύριε Τάραντ, να μιλήσουμε και για τα άλλα τμήματα πριν δώσουμε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής. Ο κύριος Τάραντ, παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ανάλυση μου δεν θα είναι τόσο μακροσκελής. Διότι το, η δική μου ευθύνη για τη, για, τη δαπάνη, την οικονομική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ μικρότερη από αυτή του κυρίου Γκάιερ. Ήθελα λίγα σχόλια να κάνω μόνο σε αυτό το στάδιο, το προκαταρκτικό. Σημειώνω ότι το Συμβούλιο ανησυχεί για τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά δεν φτάνει, δεν επιτυχάνει το στόχο μείωσης προσωπικού του 5%. Και χαίρομαι, γιατί ακούσαμε από τους ε, κυρίους και τις κυρίες σας όλοι, Βίλαντ και Γενικό Γραμματέα, για το τι συμβαίνει. Και αυτά που ακούσαμε με πείθουν εμένα ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Στη συνέχεια υπάρχει μια κάποια σύγχυση για την Επιτροπή των Περιφερειών και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ή τις Οικονομικές και Κοινωνικές Επιτροπές στη σύσταση αυτών. Φαίνεται ότι ο Γενικός Γραμματέας κ. Βέλε έχει καθησυχάσει και διαβεβαιώσει τις Επιτροπές ότι δηλαδή οι προηγούμενες συμφωνίες θα τηρηθούν. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να επαναλάβω ότι πιστεύω ότι σε βάθος χρόνου οι επιτροπές αυτές και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσαν να συνεργαστούν περισσότερο και να μοιραστούν πλήρως τις υποστηρικτικές τους λειτουργίες και υπηρεσίες και να τελειώσει αυτός ο πόλεμος με ε, καταμέτρηση θυμάτων από τη μία και την άλλη μεριά. Υπάρχει ένα θέμα με το δικαστήριο, διότι οι περικοπές του Συμβουλίου είναι αρκετά μεγάλες εδώ. Και κατά την άποψή μου, εάν συμφωνούν και οι συνάδελφοι εδώ στην Επιτροπή, καλό θα είναι να διορθώσουμε αυτή την προσέγγιση είναι ιδιαίτερος γελίο το Συμβούλιο να επικρίνει το δικαστήριο για το κόστος λειτουργίας τους, ενώ όλοι θυμόμαστε ότι το δικαστήριο ζήτησε 7 περισσότερους ή 12 περισσότερους δικαστές. Αλλά το Συμβούλιο είναι αυτό που αποφάσισε ότι κάθε κράτος μέλος πρέπει να έχει αντικαταστάτη. Επομένως η κατάσταση αυτή φέρνει όλους σε δύσκολη θέση κατά την άποψή μου. Και υπάρχει και ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί, που το έθεσαν οι πολύ καλοί συνάδελφοι στην ΑΦΕΤ, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Και ο κύριος Μπρόκ, ο κύριος Γκουαλτιέρη και ο κύριος Φερχόφστατ, τα, τα βαρέων βαρών μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με τη Βρετανική Δημοσιογραφία πρόταση να υπάρξει σημαντικό αποθεματικό για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, για τον προπολογισμό της υπηρεσίας αυτής. Και παρόλο που καταλαβαίνω τη συλλογιστική τους, Νομίζω ότι εμείς εδώ στην Επιτροπή Προϋπολογισμών οφείλουμε να εργαστούμε σκληρά για να εντοπίσουμε μία πρόταση ή μία θέση η οποία να μπορεί να είναι δεκτή από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Αυτά ήθελα να πω για να τονίσω τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουμε, που εγείρονται ε, μπροστά μας κατά την άσκηση διαμόρφωσης τελικής θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εν ώψη των διαπραγματεύσεων και ας δούμε τι μπορεί να γίνει ε, στον τρίλογο, στον τριμερή διάλογο στη συνέχεια. Αυτά ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Τάραντ ο κύριος ε, Νούρισαν, ο πρώτος εγγεγραμμένος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μύρεσαν, ε, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σας πω κι εγώ κάποια σχόλια από δικής μας πλευράς. Όταν λάβαμε το σχέδιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνειδητοποιήσαμε ότι ο προπολογισμό είναι πολύ σφιχτός και μάλιστα έρχεται σε πολύ δύσκολες συνθήκες, γιατί θα πρέπει να διασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση παραδοσιακών πολιτικών της ΕΕ, κυρίως αυτές που στοχεύουν στη δημιουργία θέσης απασχόλησης και βιώσιμης ανάπτυξης. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να υπάρξουν χρήματα για την αντιμετώπιση σημαντικής και επίγουσης προσφυγικής κρίσης στην Ευρώπη. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι ο προϋπολογισμός είναι σφιχτός, το κατανοούμε αυτό, αλλά δεν καταλαβαίνουμε τι έκανε το Συμβούλιο με τις περαιτέρω περικοπές του Ιουλίου. Και αν δούμε τις περικοπές που έκανε το Συμβούλιο στον τίτλο 1α, εκεί φαίνεται ξεκάθαρα ότι αυτά δεν αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητες που συμφωνήθηκαν στην έγκριση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Το Συμβούλιο χρησιμοποιεί ε, τον προϋπολογισμό θεωρητικά για να λύσει την ε, εξίσωση μεταξύ δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και στήριξης της οικονομικής ανάπτυξης. Έτσι θα πρέπει να γίνεται. Τώρα, έχουμε και το ΕΦΣΥ και Υποτίθεται ότι πρέπει να αποκατασταθούν αυτές οι περικοπές των χρημάτων που πήγαν στο ΕΦΣΙ. και προς το 1Β, όπως είπε και ο Γενικός Εισηγητής, είδαμε το σχέδιο πληρωμών, ε, η, η περικοπή άνω του 20% του Payment Appropriations στον τίτλο 1Β είναι υπερβολικά πολλά και μας ανησυχούν. Ζήτησαμε περαιτέρω διευκρινήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το περιμένουμε αυτό στην αυριανή διοργανική σύσκεψη για τις πληρωμές. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ανάγκες πληρωμών για το προηγούμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Περιμένουμε όμως τα επιχειρησιακά προγράμματα να προχωρήσουν, να επιταχύνουν το ρυθμό εφαρμογής τους ε, την επόμενη χρονιά και άρα θα χρειαστούν περισσότερα χρήματα για πληρωμές. Άρα χρειαζόμαστε πιο ενήμερη αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, πιο καλή αξιολόγηση για τις εκτιμήσεις ε, σε σχέση με τις εκτιμήσεις που έστειλαν τα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί ο κίνδυνος που ελοχεύει είναι ο εξής. Να ε, συσσωρεύσουμε καθυστερήσεις στις πληρωμές και αν δεν είμαστε σε θέση να πληρώσουμε τους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε μειώνεται σαφέστατα η αξιοπιστία μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί και πέρα, η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Το έθιξε το θέμα ο εισηγητής και τώρα και παλαιότερα να πω ότι πρέπει να ευθυγραμμιστούμε εδώ με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έτσι όπως φαίνεται στην έκθεσή μας για την αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Λέμε σαφέστατα ότι η ανεργία των νέων υπάρχει, παραμένει εξαιρετικά υψηλή στην Ευρώπη και πρέπει να βρούμε περισσότερα μέσα για να χρηματοδοτήσουμε σχετικές πρωτοβουλίες βάσει του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Και το αναφέρω γιατί είναι σαφέστατα ότι ό,τι περιέχεται στην έκθεση του Κοινοβουλίου, συνταχθέν από τον κύριο Όλμπριχτ και την κυρία Τομά. Όλα όσα έχουν αποτελέσει τη θέση μας και τις προτεραιότητες μας στο παρελθόν πρέπει να αντικατοπτρίζονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης για την επόμενη χρονιά. Και ως προς τον τίτλο 2, είναι σαφές ότι πρέπει να αποκαταστήσουμε τις περικοπές που έκανε το Συμβούλιο και να αποκαταστήσουμε τα επίπεδα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την, των τροφίμων σε όλη την Ευρώπη και ως προς τη δέσμη μέτρων που πρότεινε ο Επίτροπος Χόγκαν την περασμένη εβδομάδα. Μιλούμε για τα 500 εκατομμύρια ευρώ και το γάλα βεβαίως το στηρίζω, αλλά να καταλάβουμε την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Μπρέζα μπορεί να μας διαφωτίσει ποιος θα είναι ακριβώς ο αντίκτυπος στον προϋπολογισμό για την επόμενη χρονιά. Για τον τίτλο 3, οι οροφές είναι πολύ χαμηλές. Αυτό το ξέρουμε και το έχουμε πει και το έχουμε βάλει στην αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου στη σχετική έκθεση. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της αναθεώρησης του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτά είχα να πω ε, ως προκαταρκτικές παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ο κύριος Μάνκα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τον Γιένς, με την ανάλυση δηλαδή του κυρίου Γιένς Γκάιερ οι περικοπές του Συμβουλίου για το 2017 δεν είναι τόσο μεγάλες όσο τις προηγούμενες χρονιές, αυτό είναι αληθές. Ορισμένες όμως από τις περικοπές θα ε, το κάνουν πολύ δύσκολο για μας. Δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους προτεραιότητάς μας. Για παράδειγμα, η Ευρώπη το 2020 είναι μια πρωτοβουλία που μοιράζεται από εκείνο το Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο. Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και αυτό θα είναι θέμα. Ε, όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα αντιμετωπίσουν περικοπές και αυτό θα έχει αντίκτυπο στην απασχόληση. Εάν το Συμβούλιο δηλαδή κάνει περικοπές στους τομείς που είναι προτεραιότητα για εμάς, τότε θα πρέπει να μπορέσουμε να δούμε τον αντίκτυπο ε, στους τομείς προτεραιότητας και στην απασχόληση. Για παράδειγμα, πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Ήδη από πέρσι, ορισμένα κρατημέλη μας έλεγαν ότι η πρωτοβουλία για την απασχόληση των ε, νέων αποτελούσε εκοφαντική επιτυχία στις ε, εκάστοτε χώρες και το 80% των νέων που είχαν αξιοποιήσει αυτή την πρωτοβουλία συνέχιζαν να έχουν ε, θέση απασχόλησης ακόμα και μετά τη λήξη του προγράμματος. Είναι λοιπόν μια τρομακτική επιτυχία. Θέλουμε να γίνει αξιολόγηση αυτού του ε, project φέτος. Ξέραμε ότι ήταν καταπληκτικό. Ορισμένες χώρες ήδη βλέπουν την επιτυχία όμως δεν έχουμε μία επίσημη αξιολόγηση, έκθεση προόδου για την εφαρμογή του προγράμματος επιτάπητος. Και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε υιοθετήσει τη σωστή ε, διοικητική προσέγγιση ε, για το συγκεκριμένο αυτό πρόγραμμα. Σε ό,τι αφορά ε, τα άλλα θεσμικά όργανα, ο κύριος Τάραντ αναφέρθηκε και περιέγραψε την πρόθεση μείωσης του προσωπικού κατά 1% κάθε χρόνο αθρηστικά. Οι μειώσεις αυτές να φτάσουν στο 5%. Οφείλουμε όμως να απευθύνουμε το εξή ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν κάνουν περικοπές μειώνοντας τον αριθμό των μόνιμων ε, υπαλλήλων διερμηνέων και τους αντικαθιστούν με freelance διερμηνείς, θα στοιχήσει αυτό το ίδιο με ελεύθερους επαγγελματίες διερμηνείς και όχι με μόνιμους υπαλλήλους. Επομένως, πού είναι η εξοικονόμηση και η αποταμίευση εδώ. Σαφέστατα πρέπει να υπάρχουν αποθέματα στο προϋπολογισμό. Έχω και κάποια άλλα σχόλια να κάνω, θα πάρω το λόγο αργότερα. Όμως, για τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επιτρέψτε μου να πω τα εξής. Αυτή τη στιγμή ε, δαπανούμε χρήματα για να ενισχύσουμε την ασφάλεια των κτηρίων. Και ναι, είναι σημαντικό πράγμα η ασφάλεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προκαλεί κατάπληξη όμως το γεγονός ότι ξαφνικά βρίσκουμε εκατομμύρια για την ασφάλεια του κτηρίου. Όταν όμως τα χρειαζόμασταν προηγουμένως για άλλα πράγματα και για άλλες προτεραιότητες δεν τα βρίσκαμε. Πού ήταν κρυμμένα είναι μια παρατηρήση που αξίζει να γίνει. Άλλωστε, ο πληθωρισμός θα είναι τελικά πολύ ε, χαμηλότερος από τις προβλέψεις της διοίκησης. Η διοίκηση έχει βάλει πολύ μεγάλο συντελεστή ε, προβλέποντας ε, διακοιμάσεις στον προπολογισμό οι οποίες τελικά δεν υλοποιούνται και αυτό σημαίνει ότι μετά προκύπτουν δεκάδες εκατομμυρίων ευρώ να αιωρούνται εδώ και εκεί στον προπολογισμό και να μπορεί κανείς να τα χρησιμοποιήσει κατά βούληση. Να είμαστε σαφείς και να χρησιμοποιήσουμε ε, αληθινά νούμερα ε, όταν προβλέπουμε ε, τιμές, για παράδειγμα, του κόστους της ενέργειας, να μην βάζουμε φανταστικά νούμερα που έχουμε επινοήσει, αλλά πολύ πιο ρεαλιστικά. Ε, στο ψήφισμά μας είπαμε ότι ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες και όχι επί τη βάση αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία να, είναι μια ευκαιρία να συντάξουμε προϋπολογισμό ε, με βάση τις πραγματικές ανάγκες και όχι με φανταστικά νούμερα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νεγκρέσκου. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ειλικρίνειά του. Ταυτόχρονα να παρατηρήσω ότι από ό,τι φαίνεται εμείς εγκαταλείπουμε τις θέσεις μας και δεχόμαστε αδιαμαρτύρητα τις προτεραιότητες του Συμβουλίου και τις περικοπές του. Και ξεχνάμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μία πρόταση με περικοπές, αλλά χωρίς νέες προτεραιότητες και χωρίς προσδοκίες θα έλεγα. Η συζήτηση λοιπόν για τον προϋπολογισμό και λόγω του Brexit γίνεται με πολύ κακό τρόπο. Εγώ θα ήθελα να εμείνω λίγο στις προτεραιότητές μας. Δεν τις βλέπω λοιπόν τις προτεραιότητες ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως επίσης ούτε και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να γίνει μια πιο συγκεκριμένη συζήτηση για το τι πρέπει να κάνει ο προϋπολογισμός. Κάθε χρόνο, όπως είπε ο κ. Μάνκερ, Κάθε χρόνο κάνουμε κάποιες επιμέρους ρυθμίσεις και στο τέλος ε, οι επιμέρους ρυθμίσεις δεν μας λύνουν το πρόβλημα. Εμείς συζητάμε τα θέματα αυτά με πολύ κόσμο και στις εκλογικές μας περιφέρειες και ο κόσμος ρωτάει πού πάνε τα χρήματα, ποια είναι τα συγκεκριμένα αποτελέσματα της, ε, των πιστώσεων που δαπανώνται. Ο προϋπολογισμός είναι πολύ μεγάλο πράγμα, είναι πάρα πολλές οι επιμέρους γραμμές και τίτλοι αλλά είναι πολύ δύσκολο να δούμε ε, ποια είναι τα αποτελέσματα. Για να δούμε τα αποτελέσματα πρέπει να δούμε τι θέλουμε, τι προσδοκίες έχουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίζει παιχνίδι και κλεισμένων των θυρών. Εξωτερικοποιεί σε εισαγωγικά τον προϋπολογισμό σιγά σιγά. Και σύν της άλλης δεν ξέρει τίποτα και για το Συμβούλιο και τι κάνει το Συμβούλιο και κυρίως τι θέλει το Συμβούλιο. Εμείς αναφερθήκαμε στην πρωτοβουλία για τους νέους, σαν παράδειγμα, την ανεργία των νέων. Βλέπουμε τι γίνεται. Και έχω μία ερώτηση εδώ σε σχέση και με τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Εμείς δεν βλέπουμε πού είναι τα αποτελέσματα των προπαρασκευαστικών δράσεων. Ε, είχαμε κάποιες δράσεις εδώ και δύο χρόνια, εγκρίνει, ψηφίσαμε για αυτές, Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα, δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Έγινε και τροπολογία στον προϋπολογισμό, αλλά δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. Η Επιτροπή εφαρμόζει και η Επιτροπή αποφασίζει αν θα εφαρμόσει και με ποιο τρόπο θα εφαρμόσει. Νομίζω λοιπόν ότι η συζήτηση που κάνουμε για τον προϋπολογισμό σήμερα είναι μια πάρα πολύ σημαντική πια συζήτηση, έχουμε φτάσει στα όρια και θα ήθελα να γίνει μια συζήτηση ευρύτερη και με την Επιτροπή και ανάμεσα στις πολιτικές ομάδες έτσι ώστε να δείξουμε και στους εκλογείς μας ότι κάτι κάνουμε, κάτι συζητάμε επιτέλους. Και το κέντρο παρακαλώ, όχι μόνο αριστερά και δεξιά λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Τομά έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον συνάδελφο τον κύριο Γκάιερ για αυτή την πρώτη λεπτομερή παρουσίαση. Συμφωνώ με τις γενικές γραμμές, αλλά ανησυχώ ταυτόχρονα, γιατί πράγματι, όπως είπε ο συνάδελφος Νεγκρέσκου, παρά το Brexit, παρά τις διαδοχικές κρίσεις, έχουμε την αίσθηση ότι σε δημοσιονομικό επίπεδο, και δυστυχώς όχι μόνο εκεί, παραμένουμε στο να μην βλέπουμε ποια είναι η κατάσταση. Αρνούμεθα να δούμε την πραγματικότητα της θέσης του Συμβουλίου σε δημοσιονομικό επίπεδο. Τελικά, business as usual. Αν συνεχίσουμε εμείς να έχουμε νέες απαιτήσει δαπάνες, νέα έσοδα, ε, στην ουσία απεκδίουμε τον Πέτρο για να ενδύσουμε τον Παύλο δεν είμαστε σε καμία περίπτωση στο ύψος των περιστάσεων. Δεν είμαστε σε καμία περίπτωση έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια αυτό που λέω δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. Θα σας το δείξω με συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Στο 1α. Το θέμα της αποκατάστασης ε, των ποσών αυτών σχετικά με τις περικοπές που έχουν γίνει εννοώ είναι σημαντικό για να επανέλθω σε αυτά που είπε ο Γένς, η, η πιλωτική δράση για την άμυνα είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε επί της ουσίας. Ας υποθέσουμε ότι επί της ουσίας συμφωνούμε. Τότε στην συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το Κοινοβούλιο έχει ανακοινώσει μια ξεκάθαρη θέση με την ψήφο του για την αναθεώρηση του MFF, του δημοσιονομικού πλαισίου, λέγοντας ότι δεν μπορεί να υπάρχουν πλέον νέες δαπάνες εάν δεν υπάρχουν νέα έσοδα ή να υπάρξει μια σωστή στόχευση του στόχου στον οποίο ε, θα προοριστούν τα χρήματα αυτά. Λοιπόν, πάνω σε αυτό πρέπει να είμαστε απόλυτοι και θα πρέπει οι απαιτήσει τις οποίες έχουμε για την δημοσιονομική υπευθυνοποίηση να γίνουν σεβαστές και να υιοθετηθούν πλήρως από το Συμβούλιο για το 1α πάντα, έχουμε το θέμα της απασχόλησης για τους νέους και εδώ θα ήθελα να εκφράσω την οργή μου. Ξεκινάμε από μια βασική αρχή. Έχουμε την δυνατότητα να περικόψουμε μια πρωτοβουλία εάν δεν υπάρχει αξιολόγηση της Επιτροπής. Αυτή είναι μια αμφισβητούμενη αρχή βέβαια γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις η δράση συνεχίζεται μέχρι την αξιολόγηση και αν είναι κακή η αξιολόγηση το κόβουμε. Τώρα εδώ ξεκινάμε κάτι. Καλό είναι αυτό, κακό είναι αυτό. Όχι, κόβουμε τα χρήματα εκ των προτέρων χωρίς συζήτηση. Αυτό σε επίπεδο αρχής το βρίσκω ε, πραγματικά παράδεκτο. Και τι περιμένει επιτέλους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας δώσει την αξιολόγησή της. Είναι αρκετά πρακτικό να καθυστερεί κανείς τις αξιολογήσεις έτσι ώστε να καθυστερούν και να μακροημερεύουν και οι δημοσιονομικές περικοπές. Αρκετά λοιπόν, αρκετά παίζει το παιχνίδι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, περιμένουμε την αξιολόγησή της σαν τον Μεσσία. Για το ένα β εγώ θα είμαι πολύ πιο αυστηρή από το Γένς. γιατί αρνούμε να δεχθώ ε, για την πολιτική συνοχή ιδιαίτερα ότι η ευθύνη είναι αποκλειστικά των κρατών μελών. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί αν υπάρχει ένα πρόβλημα λειτουργικού προγράμματος, υπάρχει ας πούμε. Λοιπόν, υπάρχει, ας το συζητήσουμε αν μπορέσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν δεν μπορέσουμε σε εθνικό επίπεδο. Αλλά τώρα μας τραβάει τρία χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παραμένουμε σε αδιέξοδο. Διερωτώ με λοιπόν ποιον βολεύει αυτό. Και ποιον βολεύει εννοώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί τα χρήματα που δεν χρησιμοποιεί εκεί τα χρησιμοποιεί αλλού. Το λέω ξεκάθαρα εγώ δεν θέλω να διασπείρω δαιμόνια αμφιβολίας, αλλά νομίζω υπάρχει πρόβλημα και το πρόβλημα πρέπει να συζητηθεί και να κάνει κάτι επιτέλους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει μια διπλή ευθύνη εδώ. Γιατί υπάρχει επίσης και πρόβλημα σε επίπεδο συγχρηματοδότησης, το ότι υπάρχουν ε, λιγότερες δαπάνες σε επίπεδο πολιτικής συνοχής είναι ένα επιμέρους πρόβλημα. Ίσως να κάνω κάποιο λάθος εδώ, αλλά η εκκρεμότητα παραμένει. Λοιπόν, για να χορέψουμε πρέπει να είμαστε δύο, αλλά και για να μην χορέψουμε πάλι δύο πρέπει να είμαστε. Ανησυχώ λοιπόν για την περιφερειακή πολιτική, γιατί περισσότερο από την εύση η περιφερειακή πολιτική είναι η κατεξοχήν επενδυτική πολιτική της Ένωσης, η πρώτη και καλύτερη. Και αν μπλοκάρουν τα πράγματα εκεί, τότε οι επενδύσεις γενικά θα σταματήσουν. Λοιπόν, ανησυχώ. Σάρμαμα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και να πω και εγώ δύο λόγια μόνο για την ευρύτερη, γενικότερη εικόνα που διαμορφώνονται. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Γκάιερ, τον ε, εισηγητή, αλλά και τον κύριο Τάραντ Καταρχά, είναι πραγματικά εξαιρετικέ οι περιστάσει και η χρονική στιγμή την οποία διανύουμε στην παρούσα φάση και αυτό φυσικά απαιτεί και πολύ ειδικά μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν. Δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο να συμβαίνει στην πρόταση του Συμβουλίου όμω. Με το ένα από ό,τι ξέρετε, είμαστε ήδη. Έχουμε ήδη περάσει την τάφρο. Και παρόλα αυτά τα κράτη-μέλη δεν ακούν τον κόδωνα του κινδύνου που κρούμε. Και αυτό πραγματικά μας προβληματίζει. Δυστυχώ. Δυστυχώς. Κατά δεύτερον, σε ό,τι αφορά την ε, διαμόρφωση των προτεραιοτήτων. Εγώ είμαι υπέρ τη ε, διαμόρφωση τέτοιων προτεραιοτήτων και θα έπρεπε να το κάνουμε πιο πολύ στον ε, προπολογισμό της Ένωσης. Είναι σαφές για όλους μας ότι η ανάπτυξη και η απασχόληση είναι τα σημεία κλειδί. Η έρευνα και η ανάπτυξη αποτελούν τον τρόπο για να πετύχουμε όλα αυτά. Η μετανάστευση είναι κάτι το οποίο αναγκαστικά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και κατά τρίτον, το λέω αυτό συγκεκριμένα και ε, με επίγνωση ότι είμαι η φωνή της μειοψηφίας και θα διαφωνήσω με κάποιους ε, από τους προλαλήσαντες. Στο σημείο 3 βάζω την άμυνα. Δυστυχώς δεν έχει προστιθέμενη αξία, δεν είναι παραγωγικό σκέλος, αλλά είναι κάτι το οποίο στο οποίο θα επανέλθουμε. Να θυμάστε τα λόγια μου Αύγουστος 2016. Το λέω, ε, μάλλον είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να έχουμε κάνει εδώ και κάποια χρόνια ήδη. Και τουλάχιστον βλέπουμε κάτι θετικό στην πρόταση του Συμβουλίου. Είναι μικρή η αρχή, αλλά είναι μια αρχή παρόλα αυτά. Και κατά τρίτον, σε ό,τι αφορά την γενικότερη εικόνα που διαμορφώνεται, συμφωνώ απόλυτα με τον εισηγητή κύριο Γκάιερ, είναι ατυχές το γεγονός ότι το Συμβούλιο συστηματικά προσπαθεί να μειώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά θεωρώ ότι αυτό αποδεικνύει απλά το λυπηρό γεγονός ότι τα κράτη-μέλη πολύ απλά εξακολουθούν να ζουν σε άρνηση. Σε άρνηση, όπως είπε η κυρία Τωμά, πολύ εύστοχα. Αρνούνται το γεγονός ότι υπάρχει μια ε, μεγάλη κρίση, μια κρίση που απειλεί την ίδια την ύπαρξη του κόσμου στην Ευρώπη. Και θεωρώ ότι το μοναδικό αντίδοτο είναι πιο πολύ Ευρώπη. Όχι λίγο παραπάνω Ευρώπη, πολύ παραπάνω Ευρώπη. Και αυτό θα πρέπει να αποτυπωθεί και στους προϋπολογισμούς. Γιατί ο προϋπολογισμός ε, είναι ο καθρέφτης που δεν συγχωρεί, αν θέλετε, ε, του πώς έχει η κατάσταση. Και η απάντηση είναι σαφής, ξέρετε, ότι η Ευρώπη δεν ξυπνάει, δεν ε, εισακούει τις εκκλήσεις αυτές και θα πρέπει να φροντίσουμε να γίνει αυτό. Ευχαριστώ, ο κύριος Φερνάνδες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τον εισηγητή και τον σκιώδη συγητή. Ξέρετε, όλοι βρισκόμαστε στην ίδια βάρκα και συμμεριζόμαστε. Έχουμε τους ίδιους στόχους, τους ίδιους σκοπούς. Είναι η τέταρτη χρονιά του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014, 2015 2014-2015, 2016-2017 Και αυτό το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο θα έπρεπε να λειτουργεί ήδη εξαιρετικά αποτελεσματικά και απρόσκοπτα. Θα πρέπει να έχουμε κάτι υπόψη μας. Ότι ο προϋπολογισμός είναι το 1% του ΑΕΠ. Και η Επιτροπή ως προς τις πληρωμές στην πρότασή της παρουσιάζει αυτό που θέλει να ακούσει το Συμβούλιο και το Συμβούλιο ενδιαφέρεται μόνο για τα έξοδα και τις δαπάνες και όχι για τους συμβιβασμούς. Το 2017 λοιπόν που είναι το τέταρτο έτος του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου ουσιαστικά είναι το αντίστοιχο του 0,89% του ε, ΑΕΠ. και είναι λιγότερα από 10 δις ευρώ. Περικοπές. 0,89% προτείνουν από το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ότι ο προϋπολογισμός μας είναι αυτός ο λίγος για να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις που ταλανίζουν την Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Ότι δηλαδή από το 1% πάμε στο 0,89% του ακαθάριστου εγχωρίου εισοδήματος. χώρια τις περικοπές και ότι όλα αυτά πρέπει να είναι αρκετά για να επιτύχουμε τους συμβιβασμούς και τους στόχους αλλά και τις δεσμεύσεις μας. Θα πρέπει όλα να λειτουργούν απρόσκοπτα και ταχύτατα για να μπορέσουμε να ε, λειτουργήσουμε με αυτά τα χρήματα. Και αν τελικά χρειαστεί διορθωτικός, διορθωτικός προϋπολογισμός θα πρέπει να κατηγορήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί, τι σημαίνει, όταν ε, υπάρχουν διορθωτικοί προπολογισμοί για να εφαρμόσουμε τις δεσμεύσεις μας, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δοθούν περισσότερα χρήματα και χάνουμε αξιοπιστία έναντι των Ευρωπαίων πολιτών. Τελικά θα αναγκαστούμε να παρουσιάσουμε διορθωτικούς προπολογισμούς για να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας. Το βλέπω να έρχεται και θα πρέπει να το αποφύγουμε. Τώρα, ως προς τις προτεραιότητες, είναι σαφές ότι δεν θα πρέπει ο προπολογισμό να αποκλίνει από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που πραγματικά επιθυμεί ο Ευρωπαίος πολίτης. Οικονομική ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έρευνα, καινοτομία. Όλοι αυτοί είναι πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής. Ε, πρέπει να είναι παρόντες ε, ε, στον προϋπολογισμό. Καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, καταπολέμηση της ανεργίας γενικότερα. Όλα αυτά είναι προτεραιότητες για εμάς και για τους Ευρωπαίους πολίτες. Χρειαζόμαστε λύσεις. Και η πρωτοβουλία αυτή για την απασχόληση των νέων θα πρέπει να μας εξηγηθεί πού απότυχε και γιατί, ποιος έχει την ευθύνη εάν έχει αποτύχει. Και τα κράτη-μέλη έχουν ευθύνη για ε, τα στραβά. Να ξέρουμε λοιπόν ποιες είναι οι απαραίτητες προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Η ανεργία των νέων συνεχίζει να είναι διπλάσια από την ανεργία άλλων ηλικιακών ομάδων και γι' αυτό είναι αδύρυτη ανάγκη να εξευρεθούν λύσεις. Εσωτερική και εξωτερική αλληλεγγύη ζητούμε. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα. Ασφάλεια άλλη ανησυχία μεγάλη για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά όργανα της πρέπει να απεικονίσουν στον προϋπολογισμό της δράσεις προστασίας των Ευρωπαίων πολιτών. Η ασφάλεια είναι μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες στην Ευρώπη σήμερα. Σίγουρα θα βρεθεί κάποια λύση, είμαι πεπισμένος, παρά τις αποκλίνωσες απόψεις ημών ε, Συμβουλίου και Επιτροπής, όμως καλό όλους να είναι πολύ πιο φιλόδοξοι και ρεαλιστικοί συνάμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την ξεκάθαρη παρουσίασή του το Συμβούλιο είναι αντιφατικό, έχει πολλά σχήματα στο νου του, πολλά προγράμματα, αλλά δεν έχει τρόπους για την εφαρμογή τους. Και βλέπω ότι τα ποσά για τα οποία μιλάμε είναι αμεληταία για τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Παρ' όλα αυτά οι βουλήσεις των κρατών μελών είναι πλέον αποστηρωμένες. Τίθεται το θέμα των κριτηρίων σύγκλησης. Για το 1α το είπατε όλοι, είναι το θέμα της απασχόλησης των νέων. Είναι βασικό εκεί τουλάχιστον να βρούμε τη βούληση να δώσουμε λύσεις. Και βέβαια περιμένουμε την αξιολόγηση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν έχουμε την αξιολόγηση θα λύσουμε το πρόβλημα. Το θέμα της άμυνας είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το σκεφτούμε λίγο περισσότερο. Στο θέμα της άμυνας η Γαλλία είναι μαζί με την Αγγλία στην πρώτη γραμμή, το Ηνωμένο Βασίλειο. Και αν φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτό θέτει ένα πρόβλημα σε επίπεδο άμυνας και πρέπει να το σκεφτούμε. Για τα διαφορετικά ταμεία και εγώ ίδιος πρέπει να ομολογήσω ότι είμαι ιδιαιτέρως εκνευρισμένος. Γιατί τα διαφθορτικά ταμεία συνδέουν την Ευρώπη και τον πληθυσμό της. Και αν τα διαφορετικά ταμεία αυτή τη στιγμή μειώνονται, τότε και η ανάπτυξη θα μειωθεί περιπλέκουμε τα συστήματα λειτουργίας των διαφθορτικών ταμείων και αυτό αποθαρρύνει αυτούς οι οποίοι μπορεί να ωφεληθούν. Υπάρχει ένα πρόβλημα ουσίας λοιπόν, είναι το θέμα της απλοποίησης στη χορήγηση των ταμείων αυτών, των ποσών αυτών. Να δείξουμε περισσότερη εμπιστοσύνη στα κράτη-μέλη και στους τελικούς χρήστες και θα πρέπει να κάνουμε μια κατάσταση τέτοια στα πλαίσια της οποίας αυτοί που έχουν δικαίωμα στα διαφορετικά ταμεία να μην τα χρειάζονται, να μην τα ζητούν και πρέπει να υπάρξει ισορροπία ανάμεσα στις υποχρεώσεις και στις πληρωμές. Σίγουρα πρέπει να υπάρξουν κάποιες ρυθμίσεις σε επίπεδο πληρωμών, αλλά φοβάμαι ότι αν ξεφύγουμε εντελώς, ιδιαίτερα για τα διαφορετικά ταμεία θα έχουμε προβλήματα. Τώρα για το 2 για τη Γεωργία. Ήμουνα στην Επιτροπή Γεωργίας και έγινε μία μακρά συζήτηση για την πτητικότητα των τιμών. Εδώ πρέπει να γίνει πάρα πολλή δουλειά για την μελλοντική ΚΑΠ. Η μελλοντική ΚΑΠ έχει πολλές ανάγκες. Δεν μπορούμε να επαναλαμβάνονται συνεχώς ε, οι κρίσεις και εμείς να τις βλέπουμε να εξελίσσονται. Για το 4 είπε ότι θα πρέπει να αποκαταστήσουμε τις ισορροπίες, η αξιοπιστία της Ευρώπης, η στρατηγική της Ευρώπης στον κόσμο, ποια είναι, πώς εμείς θα δούμε τη Μέση Ανατολή, πώς θα δούμε τα προβλήματα ε, των υπολείπων περιοχών και η ίδια η Ευρώπη εδώ μπορεί να αμφισβητηθεί. Πρέπει λοιπόν και σαν Κοινοβούλιο και σαν Συμβούλιο να μπορέσουμε να αντιδράσουμε. Για τα υπόλοιπα τμήματα να πω ευχαριστώ στον κύριο Τάραντ γιατί ξεκαθάρισε τα πράγματα. Τα πράγματα εξελίσσονται, δεν έχω να πω πολλά. το θέμα των διερμηνέων ανάμεσα στην Περιφερειακή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το Οικονομικό και Κοινωνικό. Πρέπει να βρεθούν κάποιες συνθήκες αμοιβαιοποίησης έτσι ώστε να μπορέσουν όλα τα όργανα να εργάζονται κάτω από σωστές συνθήκες. Αυτά. Ευχαριστώ τον εισηγητή Άλμπρεχτ. Oui, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μία πολιτική παρατηρήση, επιτρέψτε μου, και μία ερώτηση να θέσω. Καταρχά, σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για τον προπολογισμό στα πλαίσια τη Επιτροπή μα, είναι τεχνική φύσεω. Ε, τώρα, μάλλον, ε, το τεχνικό σκέλος έχει ε, επισκιαστεί ουσιαστικά από το πολιτικό σκέλος. Γιατί αυτό που είπε και ο συνάδελφος είναι ότι ουσιαστικά συζητάμε κατ' ουσίαν το πρόβλημα της Ευρώπης μέσω του προπολογισμού. Γιατί σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό σκέλος είναι σαφές ότι το 1% του ακαθάριστου ε, εθνικού εισοδήματος δεν μπορεί να επιλύσει τα προβλήματα όλων των κρατών μελών. Θα πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα αυτό προ όλου. Το 1% δεν θα λύσει τίποτα. Η ανεργία αποτελεί πρόβλημα, για παράδειγμα. Με 1% για 28 κράτη-μέλη τι θα πετύχουμε. Εδώ λοιπόν χρειάζεται μια ξεκάθαρη συζήτηση. Τι εξυπηρετεί ευρωπαϊκό προπολογισμό. Αποτελεί κίνητρο. Δυναμητίζει καταστάσει Τι σκοπό εξυπηρετεί γιατί πλασάρεται ω εργαλείο που θα επιλύσει όλα τα προβλήματα. Δεν επιλύει τα προβλήματα όμω όλα. Άρα ας μην ε, το παρουσιάζουμε έτσι. Αν ε, λοιπόν έτσι είναι τα πράγματα, γιατί το χρειαζόμαστε τον προπολογισμό συμβολικό, είναι αυτό το περικόψουμε όσο θέλουμε. Δεν αριθεύει όμω αυτό. Και ουσιαστικά νομίζω ότι συζητάμε την ουσία που εξυπηρετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τι θέλουμε να πετύχουμε από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, τι θέλουμε να πετύχουμε με τι δραστηριότητέ μα. Πιστεύουμε, νομίζω ότι ένα τμήμα ημών πιστεύει, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, το ότι είμαστε μαζί, το ότι εξυπηρετούμε τα ατομικά μα συμφέροντα. Τα κράτη-μέλη τι λένε, ότι ας συνεχίσουμε όπως ε, ε συνεχίζαμε ως τώρα, ας μην αλλάξει τίποτα. Αλλά νομίζω ότι αντιμετωπίσαμε διάφορα ακαθόδε ζητήματα το Brexit και το θέμα της άμυνας. Έχουμε πολλά μεγάλα ζητήματα στο θέμα της άμυνας και εμείς κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε αυτά που βρίσκονται μπροστά στα μάτια μας. Κατά δεύτερον, Μία ερώτηση προς τον κύριο Γκάιερ. Σας συγχαίρω γιατί είστε πολύ ευγενικός και τα διαμορφώνετε αυτά με πολύ ευγενικό τρόπο κυρίως, αλλά νομίζω ότι ακολουθείτε μια πιο ομή προσέγγιση στην ουσία. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει το ερώτημα που έχω να θέσω και νομίζω ότι συμφωνεί μαζί μου και η κυρία Τωμά. Τι πρόταση έχετε να κάνετε για να υπάρξει ο σύνδεσμο μεταξύ του προπολογισμού του 2017 και της ενδιάμεσης αναθεώρησης γιατί ιδιαίτερα οι σοσιαλιστές συνάδελφοι τονίζουν αυτή τη σύνδεση. Άρα, ποια πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι η σύνδεση αυτή. Είναι η αιρεσιμότητα αυτός ο σύνδεσμος ή κάτι άλλο. Και ένα τρίτο θέμα, τεχνικό. Σε ό,τι αφορά την ε, πολιτική συνοχή στην περιφερειακή πολιτική, έχουμε το εξή πρόβλημα. Γιατί στην Επιτροπή Προπολογισμού θα πρέπει να έχουμε σαφή ενημέρωση για την περιφερειακή πολιτική από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί λοιπόν υπάρχει αυτή η καθυστέρηση γιατί θεωρώ ότι αυτή η καθυστέρηση οφείλεται σε διάφορα στοιχεία και θα πρέπει να μας ενημερώσουν ξεκάθαρα. Γιατί η του χρόνου, συμφωνώ απόλυτα, θα έχουμε προβλήματα με την ίδια την πολιτική συνοχή. Ποιο φταίει, τι συμβαίνει, γιατί έχουμε όλοι μας καθυστερήσει τόσο και στις πληρωμές και στην κατάθεση των λειτουργικών προγραμμάτων. Τα οι πράξεις κατά εξουσιοδότηση για την αριθμότητα εξάντα και αυτές δεν είναι έτοιμες. Γιατί? Για το backlog, για παράδειγμα, το οποίο μας είχαν, είχαν υποσχεθεί ότι θα μειωθεί. Όντως. Τώρα είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Το πρόβλημα όμω είναι ότι δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Γιατί αν, έχουν ξεκινήσει, αν ξεκινήσουν τα προγράμματα, θα ξεκινήσουν οι πληρωμέ. Και το backlog για το επόμενο διάστημα θα είναι μεγάλο. Άρα δεν ε, υπάρχει backload γιατί δεν έχουν ξεκινήσει οι πληρωμές. Τι θα γίνει σε δύο χρόνια όμως. Παίρνουμε χρήματα από τα περασμένα έτη, ε, χρησιμοποιούμε τα ταμεία εκτακτή ανάγκη. Τι θα γίνει σε τελική ανάλυση όμως με την ε, πολιτική συνοχή. Ενδεχομένω κάποιοι να υποστηρίξουν ότι είναι άχρηστη γιατί πρόκειται για διανομή χρημάτων, γιατί δεν είναι επενδύσεις, γιατί δεν θα έχει αποτέλεσμα. Άρα θεωρώ ότι καταρχάς θα πρέπει να αναλύσουμε σωστά την κατάσταση όσο έχει. Τι συμβαίνει, πού είναι τα προβλήματα, πώς μπορούμε να τα επιλύσουμε. Θεωρώ ότι δεν ε, μπορούμε να περιοριστούμε στο τεχνικό σκέλος. Θα πρέπει να επιστρέψουμε σε μεγαλύτερο βάθος. Θα πρέπει να γίνει μια πιο σοβαρή συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα μπορέσουμε να το αποφύγουμε αυτό και στα πλαίσια της συζήτηση για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Γιατί στο θεωρώ ότι η γενικότερη πολιτική μάλλον ε, συντείνει προς την ε, μείωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαραγκάλ. Ευχαριστώ. Ναι, Νομίζω ότι ακούστηκαν τα περισσότερα. Λίγα είναι αυτά τα οποία έχω να πω. Οι δυσκολίες μπροστά μας είναι πάρα πολλές. Πρέπει για μια ακόμη φορά να δώσουμε μια μάχη για τα ψηλά σε εισαγωγικά. Μια συζήτηση για τις λεπτομέρειες μετά από τις προκλήσεις του Συμβουλίου. Δεν θα πρέπει να εγκαταλείψουμε τις αρχές μας, δεν πρέπει να αποκλίνουμε από τις αρχές μας. Το 17 είναι ο πρώτος προϋπολογισμός μετά την αναθεώρηση, δεν πρέπει να το αγνοήσουμε αυτό. Έχουμε αν θέλετε μια νέα βάση εκκίνησης εδώ. Δεν μπορούμε σαν κοινοβούλιο να εγκαταλείψουμε τη θέση αυτή και θα πρέπει να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη συνεκτικότητα και σε σχέση με τις κατευθυντήριες ε, του 17 και σε σχέση με την ενδιάμεση αναθεώρηση. Νομίζω ότι αυτά είναι τα δύο βασικά σημεία από τα οποία θα ξεκινήσουμε. Ευχαριστούμε κύριε Γκέγερ για το working document. Είναι πραγματικά αντικειμενικό, ε, πλήρες θα έλεγα, μας δείχνει πως είναι η κατάσταση, δεν έχω τίποτα να πω. Δείχνει το μέγεθος της δυσκολίας που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Δεν ξέρω αν για μια ακόμη φορά θα πρέπει να υπάρξει μια κατελάχιστον συμφωνία όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Στην ουσία όμως με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιούμε και τις δυνατότητες μας και όχι μόνο το πρόβλημα. Νομίζω ότι μετά από μια ανάγνωση του εγγράφου εργασίας είναι πάρα πολύ δύσκολο να εντοπίσει κανείς ένα ξεκάθαρο ε, μήνυμα, μια σαφέστατη πολιτική προοπτική, μια στρατηγική ευρωπαϊκή στις προτάσεις του Συμβουλίου. Μόνο περικοπές. Και στην ουσία είναι θέματα τα οποία επαφίενται στα συγκεκριμένα εσωτερικά συστήματα ισορροπιών του κάθε κράτους μέλους. Δεν έχουμε με μια πραγματικά ευρωπαϊκή πολιτική και για τις πληρωμές αυτό το οποίο γίνεται είναι να επιβεβαιώσουμε ουσιαστικά με συμβολεογραφικό τρόπο τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη, κάποια κράτη-μέλη για να εφαρμόσουν τα προγράμματα αυτά τα οποία καλούνται να χρηματοδοτήσουμε. Και αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και σήμερα και στο μέλλον σε σχέση με τις πληρωμές πρέπει λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι ισορροπίες οι οποίες κρατούν αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο και να μην αγνοούνται τόσο πολύ οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι απαράδεκτο η χρηματοδότηση της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας να γίνεται εις βάρος της πολιτικής γειτονίας, της πολιτικής εγκύτητας και της πολιτικής ανάπτυξης. Δεν είναι εναλλακτικέ οι πολιτικές αυτές. Δεν παίρνουμε από τη μία για να δώσουμε από την άλλη, δεν κόβουμε από τη μία για να ενισχύσουμε την άλλη. Γι' αυτό λοιπόν <clears throat> θα προσπαθήσουμε και μέσω των τροπολογιών μας να υπερασπιστούμε κάπως κάποια προγράμματα όπως το Horizon 2020 κτλ να αντέξουν ε, και να χαρακτηρίσουν ε, το ε, πολιετές δημοσιονομικό μέχρι το 20. Οφείλουμε λοιπόν εμείς να αποκαταστήσουμε τις περισσότερες περικοπές, οφείλουμε να ενισχύσουμε τις προσπάθειες που γίνονται για το ΕΦΣΥ, να δούμε πώς θα πετύχουμε ακριβώς την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων που είναι κατεξοχήν ευρωπαϊκά και τα οποία υφίστανται συνεχώς τις επιθέσεις, τις επιθέσεις του Συμβουλίου. Η Κύπρος, η Γαλλία, η Ελλάδα, ακριβώς όπως έχει γίνει μέχρι τώρα στις συζητήσεις μας ακολουθούν συγκεκριμένες τάσεις και βλέπουμε απαράδεκτο χώρες όπως η Ισπανία να μην συμμετέχουν στη συζήτηση αυτή. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι προτάσεις του Συμβουλίου δημιουργούν προβλήματα και υπονομεύουν την λειτουργικότητα πάρα πολλών προγραμμάτων του Συμβουλίου επιτίθενται ακριβώς με το άλοθη της μείωσης του διοικητικού κόστους κάθε φορά. Αυτό δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία των προγραμμάτων αυτών. Δεν είναι μόνο τεχνικό το θέμα, είναι λειτουργικό κυρίως. Και στην ουσία περικόπτουν πολιτικές υψηλού ευρωπαϊκού ε, περιεχομένου, μειώνουν τις δυνατότητες χρήσης της ευελιξίας, μετά μάλιστα και από θέσει τις οποίες έχουν οι ίδιες αυτές χώρες υπερψηφίσει στα πλαίσια του νέου δημοσιονομικού προγράμματος. Θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το πολιτικό περιεχόμενο της συζήτησης αυτής, αυξάνοντας και τα κριτήρια και τις προτεραιότητες ε, τις οποίες έχει το κοινοβούλιο αυτό και μετατρέποντας τις πολιτικές αυτές προτεραιότητες σε δημοσιονομική γλώσσα, μεταφράζοντάς τις σε δημοσιονομική γλώσσα. Ελπίζω λοιπόν ότι οι τροπολογίες μας θα βοηθήσουν και τον εισηγητή και τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες έτσι ώστε να καταλήξουμε τελικά σε μια πρόταση για έναν προϋπολογισμό ευρωπαϊκό, έναν κατεπήγοντα προϋπολογισμό που να καλύπτει τις ανάγκες της Ευρώπης. Περιμένουμε λοιπόν με ανυπομονησία την πρόταση της Επιτροπής για το δημοσιονομικό το πολιετές γιατί αλλιώς φοβάμαι ότι η συζήτηση την οποία κάνουμε δεν θα έχει και ιδιαίτερο περιεχόμενο. Ευχαριστώ λέει ο πρόεδρος, ο κύριος Κόλμελ. Ευχαριστώ πρόεδρε και καταρχάς να ευχαριστήσω τους, ε, τον συνάδελφο Γκάιερ και τον συνάδελφο Ταραντ για την λεπτομερή αυτή επεξεργασία και για την πολύ σωστή παρουσίαση εδώ. Και χαίρομαι που η συζήτηση αυτή σήμερα ανέφερε σε διάφορες περιστάσεις τις εξής ε, αρχές. Χρειάζεται μία συζήτηση επί της αρχής για το τι θέλουμε να πετύχουμε με τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι μπορούμε να πετύχουμε με τον προϋπολογισμό. Γιατί αυτά είναι δύο βασικά στοιχεία. Και φυσικά πάντα υπάρχουν ελλείψει. Κανένα κράτο δεν έχει όσο χρήματα θα ήθελε να ξοδέψει και να δαπανίσει σε αυτόν τον κόσμο. Άρα το ίδιο συμβαίνει και στη δική μα την περίπτωση. Το ερώτημα λοιπόν είναι, όντω, Ποια είναι η σωστή κατεύθυνση προς την για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή που διανύει η κρίση, Όντω. Και εδώ λοιπόν διαπιστώνουμε ότι θέλουμε φυσικά όλοι μια καλύτερη Ευρώπη. Ασφαλώς. Πώς θα το πετύχουμε όμως αυτό. Με πιο πολλή Ευρώπη ή με πιο λίγη Ευρώπη για να δημιουργήσω και αυτή την αντέθεση. Εδώ λοιπόν πρόκειται για ένα θέμα αρχής όντως. Και λαμβάνοντας υπόψη τα όσα έγιναν στα πλαίσια του Brexit, δεν ε, ψήφισαν υπέρ του Brexit η Βρετανία επειδή φοβούνται ότι θα έχουμε λιγότερη Ευρώπη. Και άρα είναι σημαντικό, θεωρώ, να ξεκαθαρίσουμε το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούμε. Το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούμε εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι οι πολίτες της Ευρώπης. Τι θέλει δηλαδή ο πολίτης στην Ευρώπη. Και στην παρούσα φάση έχω έντονα την αίσθηση ότι πολλοί πολίτες δεν ε, είναι υπέρ πιο πολλή Ευρώπης. Γιατί δεν ξέρουν τι συμβαίνει αυτό. Όχι σε αφηρημένο επίπεδο, αλλά συγκεκριμένα σε επίπεδο λεπτομέρειας. Τι σημαίνει αυτό. Και έτσι ενδεχομένως θα μπορούσαμε να πείσουμε τους πολίτες να υποστηρίξουν περισσότερη Ευρώπη. Αυτό φυσικά δεν το ξέρουμε. Εγώ στην παρούσα φάση είμαι πολύ διστακτικός για το κατά πόσον ε, μπορούμε να πετύχουμε, να κάνουμε ένα βήμα πιο προς την μεγαλύτερη Ευρώπη, παίρνοντα μαζί μας και τους πολίτες. Θεωρώ ότι αυτό θα προαπαιτούσε πάρα πολύ χρόνο. Και γι' αυτό πρέπει να σας πω ότι ο προϋπολογισμός αυτός ως έχει από πλευράς ε, βασικών κατευθυντηρίων γραμμών ε, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα κράτη-μέλη στενεύονται. Δεν έχουν άλλα χρήματα και δεν θέλουν να εξοδεύσουν ενδεχομένω άλλα χρήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εμεί θα πρέπει να βγούμε να διαφημίσουμε ότι αξίζει τον κόπο να επενδύσουμε πιο πολλά χρήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά χρειαζόμαστε προς την κατεύθυνση αυτή συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τα θέματα της αναπτύξης μιας κοινή ευρωπαϊκής άμυνας. Μου λείπουν συγκεκριμένε προτάσει. Τι θέλουμε συγκεκριμένα να συμβεί. Όσο δεν το ξέρουμε αυτό, Πώς θα κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις και πώς θα ξοδέψουμε πιο πολλά χρήματα. Και το ίδιο συμβαίνει και ακόμα χειρότερα τα πράγματα σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό και το θέμα του ασύλου. Πρώτα θα πρέπει να τεθεί ο πολιτικός στόχος και μετά θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα υλοποίηση για την επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί. Και μετά, μόνο μετά, σε τρίτη φάση διαμορφώνεται ο προπολογισμό. Έχουμε ένα πολιτικό στόχο, αλλά δεν έχουμε το πρόγραμμα υλοποίηση και παρόλα αυτά θέλουμε ε, να προβλέψουμε ποσά στον προπολογισμό. Δηλαδή, ποσά τα οποία θα υλοποιήσουν τι ακριβώ τελικά. Παρόμοια είναι η κατάσταση και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Έχουμε ένα στόχο, θέλουμε να επενδύσουμε. Αλλά μέχρι και την τελευταία στιγμή που ψηφίσαμε τον προπολογισμό, δεν ξέραμε πώ επρόκειτο να υλοποιηθεί. Και το αποτέλεσμα το βλέπουμε, δυστυχώ. Και άρα έχω να πω το εξή. Αυτή η συζήτηση επί τη αρχή για το πώ θα πετύχουμε μια καλύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι απαραίτητο, καταπήγον. Γιατί ο προπολογισμό κάθε κρατική ε, δομή και τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα ίδια προβλήματα, αλλά θα πρέπει να πούμε ξεκαθαρά το τι θέλουμε να πετύχουμε. Σε ό,τι αφορά την περικοπή των πληρωμών, μπορεί να αποτελεί ένα κομψό μέσο για τα κρατημέλη στην παρούσα φάση, αλλά βλέπω ότι έχουμε μία διαφορά 23 δισεκατομμυρίων σε ό,τι αφορά την ανάληψη υποχρεώσεων των πληρωμών. Αυτό αργά ή γρήγορα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην καταληξεί σε του λογαριασμούς. Αυτά. Ευχαριστώ. Ο κ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον ε, εισηγητή και πρέπει να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τις γενικότερες γραμμές που παρουσίασε. Να πω το εξή ότι στην παρούσα φάση συνεργάζομαι με την ε, συνάδελφο Μπερέσα από πλευράς της Επιτροπής ε, Προπολογισμού ε, για το θέμα των χρηματοοικονομικών, δημοσιονομικών ικανοτήτων για την Υπέτρο. Ένα θέμα το οποίο είναι αμφιλεγόμενο και θα πρέπει να συζητηθεί. Και φυσικά Υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι βγαίνουν και λένε Μα α αντιμετωπίσουμε την πραγματική κρίση που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην παρούσα φάση, το μεταναστευτικό, όπου τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Το άρθρο 78 80 της συνθήκης, υπάρχουν και κράτη-μέλη που ζητούν να ελεγχθεί ε, η ευρωπαϊκή τάξη σε ό,τι αφορά θέματα ειρήνη κτλ. Διατείνονται λοιπόν ότι αυτά είναι πραγματικά πιεστικά ζητήματα και σε ό,τι αφορά την μείωση τη δυσπιστία, την αντιμετώπιση του λαϊκισμού και του εθνικισμού μέσω σωστών δράσεων, θεωρούν ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα μα κάνει να αναλάβουμε τι ευθύνε μα. Αλλά κοιτάξτε, εδώ ο προπολογισμό παίζει σημαντικό ρόλο και φυσικά όταν πηγαίνουμε στι εκλογικέ μα περιφέρειες βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές, ε, σε πολλέ περιπτώσει τρευλή άποψη για την ευρωπαϊκή κατάσταση, λαϊκισμό σε πολλά κράτη-μέλη, στι πρωτεύουσε που προτιμούν ασφαλώ να, τα, να σπρώξουν τις ευθύνες στο ευρωπαϊκό επίπεδο και να αποποιηθούν κάθε ευθύνη. Μιλώντας για δημοσιονομικές ικανότητες και για μέτρα βιώσιμης σταθεροποίησης, γιατί εδώ αυτός είναι ο πραγματικός στόχος σε ό,τι αφορά την Ευρωζώνη, γιατί μιλάμε για την ενιαία αγορά και το νόμισμα είναι το ευρώ και τα υπόλοιπα είναι εξαιρέσεις. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση μέσω μείωσης της δυσπιστίας και μέσω τόνωσης των βασικών αρχών του ευρωβουλίου. Και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο φυσικά να πετύχουμε το οτιδήποτε και να απαιτήσουμε το οτιδήποτε όταν έχουμε τα προβλήματα τα οποία έδειξαν και οι συγητές αλλά και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Όταν η διαχείριση και η υλοποίηση των ε, ζητημάτων αυτών στην ε, πολιτική του προϋπολογισμού αποτελούν θέματα υπό αμφισβήτηση. Να μην ε, αρχίσουμε να κατηγορούμε μεν τους δε. Και όπως είπε ο Γιάνν Ολμπριχτ, θα πρέπει θεωρώ να κάτσουμε και να ρωτηθούμε το τι γίνεται, ποιος φταίει, γιατί τα κονδύλια του ταμείου, των θετικών ταμείων δεν μπορούν να απορροφηθούν. Και θα πρέπει να κοιτάξουμε τι γίνεται και στις περιφέρειες. Διαπιστώνουμε ότι Ουσιαστικά θα έπρεπε να έχουμε πιο πολλά μέσα για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, αλλά έχουμε προβλήματα εφαρμογής, υλοποίηση. Ποιο είναι υπεύθυνο εδώ. Είμαστε πλέον τόσοι, τόσο περίπλοκοι στους κανονισμούς μας που δεν μας καταλαβαίνει κανείς και δεν καταλαβαίνει και τα κρατημέλη και τα επιβαρύνουμε υπερβολικά ή μήπως τα κρατημέλη παίζουν ένα παιχνίδι μεταξύ θεσμικών επιπέδων και θα πρέπει να αναλυθούν ε, να, να ληφθούν μέτρα σε πολλά επίπεδα. Γιατί αν στην τελική ανάλυση του τέλος τη δημοσιονομικής περίοδου δεν έχουν δαπανηθεί τα ποσά αυτά, δεν έχουν καταφέρει τα κάτι μέλη να εφαρμόσουν τα προγράμματα αυτά ή για παράδειγμα στην πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, σε τελική ανάλυση δεν πετύχουμε αυτό που θέλαμε να πετύχουμε και είχαμε θέσει ως στόχο, θα πληχθεί και η δική μας ε, η φήμη και το δικό μας το κύρος είτε έχουμε συμμετέχει άμεσα είτε μόνο έμεσα στην όλη αυτή τη διαδικασία και να το τονίσω, αν και είναι για γέλια, ότι στην εφαρμογή της μεταρρύθμισης για τα γεωργικά ζητήματα, όπως είπε ο συνάδελφος Ντενανό, να αναφέρω και εγώ την πτυτικότητα των τιμών, θα πρέπει να κοιτάξουμε και τα θέματα ε, και τη σχηματισμού καρτέλ σε όλη την αλυσίδα ε, των τροφίμων και διαπιστώνουμε ότι στην παρούσα φάση πάνω από τρία τέταρτα, και έχω ακριβή αριθμητικά στοιχεία να σας πω, πάνω από τρία τέταρτα των εισοδημάτων και του κέρδους εξαρτάται από τις ε, άμεσες πληρωμές από τις Βρυξέλλες. Και όσο πιο μεγάλη είναι η κρίση και τόσο πιο πολύ εξαρτώμαστε στα δίκτυα ασφαλείας, τόσο πιο, πολύ, τόσο πιο μεγάλο είναι το ποσοστό αυτό, να μην το ξεχάσουμε αυτό απειλήσαμε να απορρίσουμε τις ε, πράξεις κατά εξουσιοδότηση στην τελευταία μεταρρύθμιση των γεωργικών ζητημάτων. Και στι κατευθυντήριες γραμμές τι οποίες συμφωνήσαμε αναφέρεται ότι υπάρχουν ε, ποσά, ότι υπάρχουν ε, μέσα και για παράδειγμα για την προστασία του περιβάλλοντος. Εξαιρετικό παράδειγμα. Το δέντρο αποτελεί ένα κομμάτι του τοπίου δεν μπορεί να κοπεί. Γένσε, γελάς. Αλλά τι σημαίνει στην πράξη όλες αυτές οι επιδιογραφές Δεν υπάρχουν ακριβείς ε, αναφορές κατά πόσον γίνεται η μέτρηση, για παράδειγμα, στην αρχή του έτους ε, ή κατά πόσον ε, γίνεται η μέτρηση στα τέλη ενός έτους. Γιατί φυσικά αναπτύσσεται το δέντρο. Και πώς γίνεται η μέτρηση, πώς την μετρούν, πώς μετρούν το ύψος του δέντρου ή διάφορες επιχειρήσεις. Και αυτό φυσικά ισχύει για πάρα πολλά άλλα ζητήματα, όπου δεν υπάρχει απαραίτητα σωστή κατανόηση από όλου. Θέλουμε λοιπόν λιγότερη νομοθεσία, αλλά πιο σαφή νομοθεσία και θα πρέπει και από δική μα πλευρά να τονίσουμε αυτό. Για να, επιβιώσουμε στην ζούγκλα αυτή των ε, νομοθετημάτων. και να θέσω και τρει φημικέ ερωτήσει. Την παράλληλη εβδομάδα αναμένουμε τις προτάσεις τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου και αναμένουμε και ένα FC2. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό θεωρώ να συνεχίσουμε σήμερα τον αγώνα. Να μην συζητάμε μόνο τις ενδεχόμενε τεχνικέ αλλαγέ, σε ό,τι αφορά την Αφρική, σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή, και εκτός του προϋπολογισμού θα πρέπει υποτίθεται να δημιουργηθούν νέοι πυλώνες χρηματοδότησης. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε από πλευράς ε, προϋπολογισμού. Έχουμε πολλές δυνατότητες, ίσως υπερβολικά πολλές δυνατότητες για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τελικά η διαχείριση γίνεται, λες και είμαστε τράπεζα, όχι ένωση. Και ουσιαστικά το βγάζουν απ' έξω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεωρώ ότι οι νέες δομές, υπό την έννοια αυτή, που θα οδηγούσαν σε παραγωνισμό του Κοινοβουλίου και παραγωνισμό των βασικών στρατηγικών ε, στόχων μας είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αποδεχτούμε. Και τώρα να περάσω στην ε, κατηγορία 4. Το είπε και ο συνάδελφος ε, ταράντσα ό,τι αφορά τα μεγάλα αποθεματικά για την έρευνα και την ανάπτυξη κτλ. Θεωρώ ότι εδώ χρειάζεται μια εντελώς καινούργια συζήτηση για τη στρατηγική κοιτώντας και τι συμβαίνει γύρω μας. Πού είναι τα πιεστικά προβλήματα. Βρισκόμαστε λοιπόν περιτριγυρισμένοι από αποτυχημένα κράτη. Η πολιτική γειτονία μας, η πολιτική ανάπτυξή μας, τι έχει πετύχει τελικά. Ή εν πάση τι δεν πέτυχε για το χύψη λόγο. Και τι θα μπορούσε να αλλάξει την κατάσταση αυτή στο μέλλον. Ιταλός, δεν θα μπορέσουμε σε καμία περίπτωση να ελέγχουμε αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας. Είναι μια συζήτηση αυτή επί της αρχής. Ούτε μπορεί να περιοριστεί φυσικά για το προπολογισμό του 2017 ενδεχομένω να περάσει και στα πλαίσια τη ενδιάμεση αναθεώρηση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μην χάσουμε άλλο χρόνο, γιατί πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση. Και το γεγονό ότι το Συμβούλιο τώρα φαίνεται ότι έχει λογικευτεί κάπω σε σχέση ε, με αυτά που στην αρχή είχαν γίνει για το Προπολογισμό το 2016, κοιτάξτε, πέρασαμε και μεγάλη κρίση το καλοκαίρι. Και δυστυχώ ε, όλα αυτά τι καταδεικνύουν, ότι χάσαμε πάρα πολύ χρόνο από το γεγονός ότι κάποια κράτη-μέλη μπλοκάριζαν τα πράγματα στο Συμβούλιο. Και θα έπρεπε να έχουν περάσει πιο νωρί η απόψη του Κοινοβουλίου. Για τις πολιτικές δράσει ένα τελευταίο πράγμα να πω. Αυτά που είπατε για τη χρηματοδότηση είναι σωστό θα πρέπει παράλληλα να έχουμε υπόψη μας ότι όταν μιλάμε για πολιτική γειτονία, όταν μιλάμε για ασφάλεια, για άμυνα, δεδομένης και την κατάσταση, κατάσταση που προέκυψε από το Brexit. Πούτιν, Έρτογαν, Τραμπ, οι πολιτικές ροές, οι πολιτικές τάσεις ε, γύρω μας. Μα υπάρχει ανάγκη λοιπόν ανάλεψης δράσης. Και δεν μπορούμε να καθόμαστε να κοιμόμαστε επί δεκαετίες. Το 79, να σας πω, ξεκίνησα για πρώτη φορά να συμμετέχω σε ευρωπαϊκές εκλογές. Ήμουν κάτω-κάτω φυσικά στην ε, λίστα. Ο κύριος Χάσελτ ήταν ο πρώτος ε, στη λίστα μου, πρώην υπουργό Άμυνα ε, στη Γερμανία και πρόεδρος του Bundestag. Μίλησε λοιπόν για την αναβίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άμυνας. Και θυμάμαι ακόμα την πρώτη συζήτηση, την πρώτη ομιλία που έκανα αντικαθιστώντας τον και προκάλεσα πραγματικά έξαλλο θυμό από όλους όσους με άκουγαν να μιλώ για Ευρωπαϊκή Άμυνα. Έχουμε χάσει τόσο πολύ χρόνο, μα τόσο πολύ χρόνο. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια κοινή στρατηγική. Και είναι ενδιαφέρον αυτό το ότι σε κάποιες συναντήσεις κρατών μελών η συζήτηση αυτή παρουσιάζεται από κάποια κράτα, από νέα κρατημέλη. Και ασφαλώς αυτό είναι μόνο ένα κομμάτι των όσων καλούμαστε να συζητήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει να καλέσουμε το Συμβούλιο να δώσει μεγαλύτερη όθεση προς την ε, κατεύθυνση αυτή. Όχι μόνο ένα πλαιτικό πρόγραμμα, αλλά και παραπάνω πράγματα, γιατί δεν έχουμε πλέον πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Παίζαμε ένα παιχνίδι όταν ήμουν μικρός, Λεγότανε πώς θα κάνουμε την Αλεπού να πεινάσει. Παιχνίδι με χαρτιά. Αυτό παιχνίδι παίζουμε και με τον προϋπολογισμό τώρα. Έχουμε όλο και λιγότερα χαρτιά στη διάθεσή μας Είδαμε τι γίνεται με το Εύση. Τα κράτη-μέλη ακολουθούν και παίζουν δικά τους παιχνίδια. Ο χώρος για κινήσεις στο εσωτερικό του προϋπολογισμού περιορίζεται όλο και περισσότερο και θα πρέπει να δώσουμε μάχη για την αποκατάσταση των περικοπών που βγήκαν από τον προϋπολογισμό ακριβώς που έγιναν ακριβώς για να τροφοδοτήσουν το εύση το στρατηγικό ταμείο. Δεύτερο σημείο, βασικό. Έχει σημασία το πώς βλέπουμε τον κόσμο όταν ο κόσμος αυτός δεν είναι αυτός που ζούμε. Εγώ διάβασα μια έκθεση ενός Ινστιτούτου για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη. Στην σελίδα 9 της έκθεσης αυτής υπάρχει μια εικόνα, μια φωτογραφία μια συγκεκριμένη απειλή στον τομέα της ασφάλειας. Όταν έχεις πάνω από 25% ανέργων από τα 15 μέχρι τα 24, τίθεται άμεσα ένα πρόβλημα ασφάλειας. Και ιδιαίτερα όταν μιλάμε για την Νότια Ευρώπη. Το θέμα αυτό της ασφάλειας Νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολήσει όλους και κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Έμεσα συνδεδεμένο με αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το ότι πιστεύουμε ότι χρειαζόμεθα περισσότερα χρήματα για τη συλλογή των δεδομένων τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούμε για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ασφαλείας. Ένα τέταρτο σημείο έχει σχέση με μια απόφαση που είχαμε πάρει στα πλαίσια της στρατηγικής Ευρώπης 2020, ότι το 20% δηλαδή του προϋπολογισμού θα πρέπει να αντιμετωπίζει και τις συνέπειες των κλιματολογικών επιπτώσεων. Το ποσοστό αυτό για του χρόνου στις προβλέψεις είναι 19,2%. 19,2% το 14 και το 15 ήμασταν μακράν του 20%, το 16 ήμασταν κοντά. 9-10 μήνες λοιπόν μετά από την COP21 στο Παρίσι, βλέπουμε ότι υπαναχωρούμε από αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε και αυτό είναι ασυγχώρητο. Εφόσον πήραμε μία απόφαση, και εφόσον δώσαμε υποσχέσεις δεν μπορούμε να υπαναχωρούμε, δεν μπορούμε να παλινοδούμε γιατί πραγματικά πρόκειται για μεγάλο πολιτικό λάθος, για να μην πω κάτι άλλο. Τζάνι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος οι περισσότεροι συνάδελφοι έδωσαν με πολλές λεπτομέρειες τις θέσεις τους. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Ελπίζω η συζήτηση να αποκτήσει πιο συγκεκριμένες πλευρές όταν κατατεθούν οι τροπολογίες για τη θέση του Συμβουλίου. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι το Συμβούλιο έχει λειτουργήσει τόσο απρογραμμάτιστα ε, αποφάσισε σε κάποιους τομείς να μην παρέμβει και να αφήσει χώρο στο Κοινοβούλιο για κάποια ευαίσθητα θέματα, τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θετικό και πρέπει να το υπογραμμίσουμε για τη θέση του Συμβουλίου. Το μοναδικό τμήμα, αν θέλετε, των θέσεων αυτών, των θέσεων του Συμβουλίου, είναι οι περικοπές των αποθεματικών για τα ειδικά μέσα. για το ΦΕΓ σαν παράδειγμα, τα ειδικά αυτά μέσα είναι αλήθεια ότι λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο από τη μια κανονική γραμμή του προϋπολογισμού. Όμως το να υπάρχει ένα αποθεματικό και εκεί βοηθά να καλυφθούν κατεπίγουσες καταστάσεις και όλο και περισσότερο έχουμε κατεπίγουσες καταστάσεις τις οποίες καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Λοιπόν δεν καταλαβαίνω ποια είναι η πρόθεση του Συμβουλίου εδώ. Ένα άλλο σημείο που πρέπει να υπογραμμίσω και πάνω στο οποίο θα πρέπει να γίνει μεγαλύτερη συζήτηση, ιδιαίτερα μετά από αυτό που συνέβη το καλοκαίρι στην Τουρκία, είναι να δούμε ποιες είναι οι θέσεις της τουρκικής κυβέρνησης σε πολλούς τομείς. Είναι απαραίτητο να βρούμε τρόπο συζήτησης εκ νέου της υποστήριξης που δίδουμε προς την Τουρκία. Εμείς δίνουμε σημαντικά ποσά προς τη χώρα αυτή, μια χώρα η οποία δεν συμπεριφέρεται με τρόπο, σε εισαγωγικά το βάζω, σωστό στις σχέσεις της με την Ένωση και στις σχέσεις της με τη διεθνή κοινότητα και εδώ αναφέρομαι και στον κοινοτικό προϋπολογισμό και στα θέματα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, γιατί η Τουρκία είναι μία από τις χώρες που παίρνει πολλά χρήματα από την BEA, BEI δηλαδή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πρέπει να δούμε λοιπόν ακριβώς τι συμβαίνει με την Τουρκία. Για τα υπόλοιπα τμήματα του προϋπολογισμού θα συμφωνήσω με τους προηγούμενους συναδέλφους και με τον εισηγητή για την Επιτροπή των Περιφερειών και για την οικονομική και κοινωνική. Θα συμφωνήσω μαζί τους ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα εξορθολογισμό του κόστους, ιδιαίτερα αφού μοιραστούμε κάποιες δραστηριότητες μαζί τους σε επίπεδο διοικητικό. Τα δύο αυτά όργανα έχω τη γνώμη ότι συνεχίζουν να παίζουν έναν ρόλο αντιιστορικό. Τι εννοώ. Εδώ και δύο χρόνια είμαι εγώ εδώ ε, και δεν έχω καταλάβει τι χρησιμότητα έχουν εν πάση περιπτώσει. Ίσως να είναι δικό μου θέμα, πάντως αντιπροσωπεύουν κάτι το οποίο ανήκει στο παρελθόν και στην ουσία είναι ένα καταφύγιο για συνταξιδιωτιωμένους πολιτικούς παλαιάς κοπής. Για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης με ανησυχεί η συνεχής αύξηση των πιστώσεων προς την υπηρεσία αυτή, χωρίς να υπάρχει μια ξεκάθαρη γραμμή και να υπάρχει μια σωστή πολιτική λειτουργίας της υπηρεσίας αυτής. Και επ' αυτού νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση. Και ένα τελευταίο σημείο και επανέρχομαι σε αυτά τα οποία είπε ο Γκάιερ για την εγγύηση για τους νέους. Στην Ιταλία νομίζω ότι Πράγματι έπαιξε θετικό ρόλο στην Ιταλία το πρόγραμμα αυτό. Προέρχεται η εντύπωση σας αυτή από ένα ταξίδι που κάνατε επί τόπου. Η ανταπόκριση που εγώ έχω, ιδιαίτερα από τη δική μου εκλογική περιφέρεια, του βορρά της Ιταλίας, ιδιαίτερα τη Λομβαρδία, ε, συζήτησα με τα κέντρα απασχόλησης, ε, συζήτησα με ανθρώπους που χρησιμοποίησαν τις δυνατότητες αυτές, και το feedback δεν είναι θετικό. Σημειώνονται πάρα πολλές δυσκολίες και στρεβλώσεις στην χρήση του μέσου αυτού και μέχρι τώρα γίνονται ανοιχτές έρευνες και ανακρίσεις όχι μόνο στη δική μου περιφέρεια αλλά κυρίως στις περιοχές του Νότου όπου το μέσο αυτό χρησιμοποιείται περισσότερο διότι είναι σαφές ότι το ποσοστό ανεργίας των νέων εκεί είναι υψηλότερο και βοηθάμε πολλούς νέους να ενταχθούν στον χώρο της εργασίας. Ρούμπιχ, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την παρουσίαση των σημείων εστίασης. Νομίζω ότι και στον προπολογισμό θα πρέπει να αναλύσουμε ποιε θα είναι οι συνέπειε του Brexit. Όχι μόνο για τον ε, προπολογισμό του Κοινοβουλίου, αλλά και τη Επιτροπή. γιατί ασφαλώς και θα έχει μακροπρόθεσμα συνέπειες. Ε, μακροπρόθεσμα θα πρέπει να αυξηθεί ο προπολογισμό, ε, γιατί σίγουρα θα ακριβίνουν τα πράγματα για το πώς θα διαπραγματευτούμε και μια έκπτωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι καθοριστικό το θέμα των ε, προσφύγων, το προσφυγικό, να το κοιτάξουμε εστιασμένα. Η Μέρκελ δήλωσε χθε ορθώς ότι έχουμε επικεντρωθεί υπερβολικά λίγο στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα μπορούσαμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και πρέπει στο μέλλον να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Δεν είναι δυνατόν 28 κράτη-μέλη να ακολουθούν μια δική τους ξεχωριστή στρατηγική και 28 φορές να κάνουν τις ίδιες δαπάνες. Νομίζω ότι για όλα τα κράτη-μέλη θα ήταν πολύ πιο φτηνό και αποτελεσματικό να διαμορφωθούν τα πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πραγματικά, επιτέλους, να πούμε ότι είμαστε κοινά, από κοινού αρμόδιοι για τα ζητήματα αυτά όπως το προσφυγικό. Δεν αφορά μόνο αυτό τις χώρες ε, Σέγγεν, είναι κοινό μας συμφέρον. Η ασφάλεια και η ασφάλιση της Ευρώπης και θα πρέπει εδώ να κοιτάξουμε και την στρατηγική συνεργασία από αστυνομίας, στρατού και εδώ στο στρατό έχουμε τη μεγάλη πρόκληση ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο ασφαλώς θα είναι πιο σωστή και αποδοτική η διαμόρφωση από το ότι να διαμορφώνεται αυτό σε εθνικό επίπεδο. Αυτό θα πρέπει να το εξηγήσουμε και στο φορολογούμενο, γιατί θεωρώ ότι η Ευρώπη σημαίνει τεράστια πλέον εκτήματα για το φορολογούμενο, αλλά θα πρέπει να τα παρουσιάσουμε αυτά τα πλέον εκτήματα. Και τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει ένα λάθος. Τα επιστημονικά αποτελέσματα και συμπεράσματα, όπως το EPRS για παράδειγμα, δεν τα έχουμε παρουσιάσει επαρκώς προς το κοινό. Και θεωρώ ότι θα πρέπει από πλευρά του Κοινοβουλίου να προωθούμε προ του ενδιαφερόμενου κύκλου πολύ πιο επιθετικά, αν θέλετε, τι πληροφορίε αυτέ. Και θα σα ε, υπενθυμίσω ότι πολλοί υπουργοί και το διαπιστώνουμε αυτό κάθε φορά όταν έχονται οι προεδρίε εδώ σε εμά. Ότι και πολλοί υπουργοί λοιπόν δεν γνωρίζουν ουσιαστικά το τι συμβαίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στις διαπραγματεύσεις ε, ε, μας ρωτούν ε, πώς, αν ρωτιόμαστε μάλλον, το πώς μπορούμε να καταφέρουμε να καταρτήσουμε μια κοινή στρατηγική από κοινού, ακόμα και αν στα πλαίσια της διαλογής δεν μπορεί η Προεδρία να κάνει σωστή συζήτηση μαζί μας. Γι' αυτό λοιπόν να επιστήσω την προσοχή σας στο εξής. Χρειαζόμαστε και μια ευκαιρία εκτενού συζήτηση όλων αυτών και με του 28 υπουργού Οικονομικών. Για να οργανώσουμε τι εργασίε μα με τέτοιο τρόπο προκειμένου να δεσμευθούν, να αισθανθούν πραγματικά δεσμευμένοι οι 28 Υπουργοί και να μα παρούν στα σοβαρά και το διάλογο μαζί μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Μπρέζα για να απαντήσει στις απαντήσεις που τέθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Παρενθετικά να πω ότι εμπιστεύομαι τον κύριο Μπρέζα και πιστεύω ότι θα μπορέσει να μας κάνει σύνοψη χωρίς να μακρηγορήσει. Πριν του δώσω όμως το λόγο θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου στον ε, εισηγητή κύριο Γκάιερ και τον κύριο Τάραντ, οι οποίοι πλαισίωσαν πολύ σωστά τη συζήτησή μας, μακροσκελή, περισσότερο χρόνο κράτησε από ό,τι είχαμε προβλέψει, αλλά ήταν μια συζήτηση πολύ επικοδομητική. Άλλωστε, Έχουμε μπροστά μας ένα, ένα προϋπολογισμό για το 1 τέταρτο του προϋπολογισμού του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου που είχε ψηφιστεί το φαινόπωρο του 2013 για πρώτη φορά και που θα εκτινόταν σε τέσσερα χρόνια. Και εμείς το, εξετάζουμε μάλλον το τελευταίο τέταρτο κομμάτι. Εν τω μεταξύ όμως έχουν μεσολαβήσει πολύ επίγουσες κρίσεις και δίνουμε απάντηση σε αυτές. Σήμερα το πρωί αναφερθήκατε επιμακρών στις απουσίες, σε ό,τι δεν θα υπάρχει στον προϋπολογισμό τούτων λεχθέντων είναι δύσκολο να μοιραστούμε τις ανησυχίες μας με τους Ευρωπαίους πολίτες, με τους συμπολίτε μας. Μπορεί ένας Ευρωπαίος πολίτης να καταλάβει τι σημαίνει αυτός ο προϋπολογισμός σε σχέση με τα διακυβεύματα. Και αν ο πολίτης δεν τον κατανοεί, τότε το ίδιο το θεσμικό όργανο κινδυνεύει, γιατί δεν αναγνωρίζεται από τους πολίτες οι οποίοι δεν το βλέπουν να έχει νομιμοποίηση. Μιλούμε για προπαρασκευαστική δράση, για παράδειγμα, στον τομέα της αμήνης, ε, πιλωτικά προγράμματα. Όλα αυτά είναι ε, στο ύψος των περιστάσεων. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με τις αμερικανικές εκλογές. Ίσως όμως ο νέος πρόεδρος ή η νέα πρόεδρος ε, ταχθεί αντίθετα με τις πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα και ενδεχομένως θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδείξει περισσότερες ικανότητες, μεγαλύτερη αυτονομία για τη δική της ασφάλεια και άμυνα. Και αν πρέπει να γίνουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις, αυτές πρέπει να γίνουν στον τομέα της έρευνας. Η Επιτροπή έχει 25 εκατομμύρια για τις προπαρασκευαστικές δράσεις, ε, κόπτει αυτές για να δώσει βάρος ενδεχομένως στην έρευνα ή αλλού. Θα πρέπει αυτά τα 25 εκατομμύρια να πάρθουν από άλλα μέσα και να αποκαταστήσουμε τη χρηματοδότηση των πιλωτικών ε, προγραμμάτων και των προπαρασκευαστικών δράσεων. Σε κάθε περίπτωση κάποιες από τις προτεραιότητες πρέπει να είναι κατανοητές από την κοινή γνώμη για να ταχθεί η κοινή γνώμη στο πλευρό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εμπιστεύουμε αυτό το εγχείρημα ε, στους ε, εισηγητές. Διαδικασίες όπως το Εράσμος για παράδειγμα, το πρόγραμμα Εράσμος είναι τρομακτικές επιτυχίες. Όταν ρωτούμε τον Ευρωπαίο πολίτη τι είναι η Ευρώπη, μας μιλάει για το Εράσμος. Εάν θέλουμε λοιπόν να παγιώσουμε την Ευρώπη θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την κοινότητα κινητικότητα των νέων και το Εράσμος μπορεί να συμβάλλει. Μένω κατάπληκτος από τις διαδικασίες που ισχύουν εντός Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ορισμένοι ε, μιλήσατε για ένα πιλωτικό πρόγραμμα για τη μαθητεία και τους μαθητευόμενους. Ίσως θα πρέπει να γίνει. Μας μπερδεύει η διαδικασία. Ε, είναι αποτρεπτική. Αυτό αποτρέπει περισσότερο καθιστά την Ευρώπη καθόλου ελκυστική. Οι 600 σελίδες είναι το εγχειρίδιο για τη διαδικασία. Ορισμένες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλουν να είναι βέβαιες ότι το ελεκτικό συνέδριο ή κάποιος άλλος δεν θα εντοπίσει κανένα λάθος και γι' αυτό έχουμε εξάντε ελέγχους και γι' αυτό έχουμε η καχυποψία πρέπει να συντάσσονται οικονομικοί κανονισμοί, κανονισμοί που να δίνουν ε, περισσότερο χώρο στο ρεαλισμό, στο να είμαστε πραγματιστές και να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Σε κάθε περίπτωση, από αύριο το πρωί που ξεκινά ο τριμερής διάλογος με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η συζήτηση αυτή θα μας επιτρέψει να προβούμε σε έναν επικοδομητικό, εξαιρετικά επικοδομητικό τριμερή διάλογο και ελπίζω να αποφύγουμε την απογοήτευση. Κύριε Πρέζα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω Θεωρώ ότι η αξιολόγηση την οποία έκανε ο Γενικός σας εισηγητής δείχνει ότι υπάρχει μια μεγάλη σύγκληση ανάμεσα στις θέσεις του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής για τα θέματα τα επιμέρους τα οποία έχουν καταρχάς οι προτεραιότητες. Η πρόταση επί του προϋπολογισμού της Επιτροπής ξεκαθάρισε τις προτεραιότητες και για την ανάπτυξη και για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών και προσφυγικών ροών από την άλλη. Νομίζω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα περιθώρια τα οποία ε, ήταν διαθέσιμα, να χρησιμοποιήσουμε επίσης και την ευελιξία που εμπεριέχεται στο δημοσιονομικό πλαίσιο και ιδιαίτερα για τα προβλήματα τα μεταναστευτικά να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα ευελιξίας και να κινητοποιήσουμε και το περιθώριο πρώτης ανάγκης. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με έναν προϋπολογισμό με ξεκάθαρες προτεραιότητες. Για τις πληρωμές, ένα θέμα το οποίο έχει τεθεί από πάρα πολλούς από εσά που πήρατε το λόγο. Υπάρχει μια ανησυχία κοινή εδώ για την εφαρμογή και την ταχύτητα εφαρμογής των νέων προγραμμάτων. Η μείωση του επίπεδου πληρωμών που προτείνεται για την πολιτική συνοχής για το 2017 αντικατοπτρίζει αν θέλετε τα στοιχεία τα οποία θεωρούμε ότι χρειάζονται με βάση τα αιτήματα των κρατών μελών και με βάση την αξιολόγηση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τα ποσοστά εφαρμογής. Αύριο άλλωστε έχουμε μια συζήτηση ειδική για τις πληρωμές και θα περάσουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Θα πρέπει όμως συλλογικά θα έλεγα να επεξεργαστούμε όλες τις πιθανότητες ανάληψης δράσης έτσι ώστε να περάσουμε το ταχύτερο δυνατόν επαναλαμβάνω ταχύτητα κρουαζιέρας να το πω, σε μια κανονική ε, μορφή λειτουργίας, ρυθμό λειτουργίας για τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Έγιναν κάποια σχόλια. Εγώ θα έτεινα εδώ να συμφωνήσω με τον Μύριο Μαρινέσκου για το ότι όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναφέρεται σωστά σε σχέση με τα προγράμματα αυτά, πιλωτικά και προπαρασκευαστικές. Νομίζω ότι υπάρχει μια συνεργασία εδώ και αρκετά χρόνια με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αξιολογούνται οι τομείς τους οποίους δραστηριοποιούμεθα. Ελέγχουμε τα αιτήματα των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Και νομίζω ότι το πράγμα λειτουργεί αρκετά καλά. Η αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γίνεται ε, δις έτος. Σίγουρα υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης, αλλά θα ήθελα να πω ότι έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα, έχουμε δημιουργήσει έναν μηχανισμό ο οποίος θα χρησιμοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα περιορισμένα είναι αλήθεια ποσά στα οποία έχουμε καταλήξει μέχρι τώρα. Τώρα για την προπαρασκευαστική δράση για την άμυνα. Προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 25 εκατομμύρια. Ε, για το 17. 80 εκατομμύρια σε τριετή προοπτική. Όλα αυτά είναι ε, πιλωτικά προγράμματα τα οποία είχαν προταθεί από το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είναι κάτι το καινούριο δηλαδή. Είναι σαφές όμως ότι υπάρχουν ε, νέες απαιτήσεις νέα περιβάλλοντα έτσι ώστε η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία να διατηρήσει τις ικανότητές της και την αυτονομία της στο νέο γεωπολιτικό ε, πρόγραμμα, πλαίσιο. Τέθηκε από τον κύριο Μουρεσάν και ένα ερώτημα για το πακέτο για τα γαλακτοκομικά. Αυτά όλα συμπεριλαμβάνονται στον διορθωτικό προϋπολογισμό, στην διορθωτική επιστολή, την οποία θα προετοιμάσουμε σε λίγες εβδομάδες. Εδώ η... Προβλέπετε ότι στα μέσα ε, Οκτωβρίου θα καταθέσουμε την πρότασή μας και νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία από κοινού θα κρίνουν αν θα πρέπει να υπάρξουν ρυθμίσεις στις πολιτικές για την ΚΑΠ για το 17. το πακέτο το οποίο είπα αφορά 500 εκατομμύρια για έκτακτα μέτρα για τον γαλακτοκομικό τομέα. Αυτό είναι κάτι το οποίο συνδέεται και με τη μείωση παραγωγής σαν διορθωτικό μέτρο στον τομέα. Στην ουσία έχουμε να κάνουμε λοιπόν με μια προσπάθεια αποκατάστασης της ισορροπίας των τιμών. <clears throat> Τι να σας πω άλλο, Ε, αν κάτι άφησα είμαι στη διάθεσή σας, ε, διμερές επίπεδο ή με άλλο τρόπο να επανέλθω. Ευχαριστώ κύριε Πρέντα. Γκέιερ, να κλείσετε παρακαλώ σύντομα αν γίνεται. Ευχαριστώ πρόεδρε, να κλείσω. Ευχαριστώ σου. Και Έχουμε καθυστερήσει πάνω από μία ώρα στο χρονοδιάγραμμα, γι' αυτό λοιπόν δεν θα μακρηγορήσω. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους. Δεν θέλω να μπω στον πειρασμό να αρχίσω να λέω την απόψέ για όλα όσα είπατε, για αυτά που είπατε εσείς κύριε Πρέζα. Ναι, όντως ε, μας λείπουν αυτά που αναφέρατε. και περιμένουμε και την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον αντικτύπο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων. Πότε θα την περιμένουμε, πότε πρέπει να την... πότε θα τη λάβουμε. Γιατί θα είναι καθοριστική η σημασία της για τις περαιτέρω συζητήσεις μας για το μέσο αυτό. Θα επηρεάσει ασφαλώς. Πείτε μας έτσι ενδεικτικά πότε μπορούμε να την ε, περιμένουμε. Και να περιοριστώ στα εξή, ε, γιατί μου έκανε και κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα ο Γιάννα Όλμπρεχτ να απαντήσω. Καταρχά, ε, συνάδελφοι, ευχαριστώ για τα κομπλιμέντα σα. Ναι, προσπάθησα να είμαι ευγενή. Μπορώ να είμαι και έτσι. Κοιτάξτε, έχω και καλή διάθεση μόλι έρχομαι από τρει εβδομάδε διακοπών στην Ιταλία, στον ήλιο. Βοηθάει και αυτό. αλλά το αργότερο αύριο στον τριμερό, στο τριμερή διάλογο είμαι βέβαιος ότι θα μου φύγει αυτή η καλή διάθεση. Θα κάτσουμε μαζί με τους εκπροσώπους του Συμβουλίου. Είχα ήδη και πολλές ανεπίσημες επαφές με τον κύριο Ούρακ, ο οποίος ε, είναι υπεύθυνο των συζητήσεων από πλευράς του Συμβουλίου. Ήταν ευχάριστη η ατμόσφαιρα θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει και αύριο, να δούμε και τις ε, πολιτικές ε, ε, καταστάσεις που οδήγησαν στις σχετικές δηλώσεις από πλευράς του Συμβουλίου. Μας ικανοποιούν λοιπόν όλα όσα έκανε το Συμβούλιο. Θα ακούσουμε λοιπόν την αιτιολόγηση αύριο τον τόσο, των όσων έγιναν από το Συμβούλιο και θεωρώ ότι δεν θα είμαστε πιο ικανοποιημένοι και πιο ε, σωστά ενημερωμένοι από αύριο. Και γι' αυτό θα μου φύγει και η καλή διάθεση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη σύνδεση αυτή, μου θέσατε το ερώτημα αυτό, σε ό,τι αφορά ε, τις διαπραγματεύσεις για το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο για τον προπολογισμό του 2017. θεωρώ ότι σωστά τα είπε ο συνάδελφος Μαριγκάλ. Καταρχάς λοιπόν, ναι, ο προπολογισμό του 2017 είναι πρώτος μετά την αναθεώρηση που συζητούμε. Και φυσικά θα πρέπει να κρίνουμε κατά πόσον, μάλλον, τι μπορούμε να περιμένουμε πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο αυτό, που ε, διαπραγματεύτησε και, και έκανε μια πρώτη συνάντηση κυκλισμένων των θυρών. Αυτό δεν μας ικανοποιεί, αφενός. Και κατά δεύτερον, να δούμε τι κάνει το Συμβούλιο. Να κάτσουμε να κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση ως συζητητές ε, για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και αντίστοιχα να προβούμε στα απαραίτητα συμπεράσματα. Και αυτό αποτελεί μία από τις εναλλακτικέ που έχουμε στην ε, διάθεσή μας. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε στην αρχή των διαπραγματεύσεων. Ξεκινήσαμε λοιπόν με τις διαπραγματεύσεις. Πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνουν διαπραγματεύσεις. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη φυσικά και όλα τα στοιχεία τα οποία θα επηρεάσουν το τι διαπραγματεύσει. Μία είναι η αξιολόγηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα στοιχεία. Και μόνο όταν θα έχουμε στη διάθεσή μα όλα αυτά τα μέσα θα μπορέσουμε να καταλήξουμε στα σωστά συμπεράσματα. Και αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε άλλωστε. Μάλιστα. Επόμενο σημείο του προπολογισμού. Διορθωτικό ε, προπολογισμό ασφάλεια των θεσμικών οργάνων. Χωσέ Μανουέλ Φερνάντε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε το διορθωτικό προπολογισμό υπαριθμών 3 του 2016, ασφάλεια των θεσμικών οργάνων. Έχουμε δύο συνεισηγητές, τον υποφαινόμενο και τον κύριο Ζεγάχ Ντεπχέ. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα το 3 για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με το τρίτο τμήμα. 15,8 δισευρώ ευρώ είναι πιστώσεις για τον τίτλο 5, διοίκηση, πρόκειται για πληρωμές. Έχουμε το 1α, είναι το υπόλοιπο από το εγχείρημα που ξεκίνησε το 2014. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε ό,τι με αφορά. Μπορούμε λοιπόν να εκφράσουμε τη συμφωνία μας για αυτά τα 15,8 εκατομμύρια, διορθώνει ο μιλητής. Προβλέπονται για την ασφάλεια 5 εκατομμύρια για τα ευρωπαϊκά σχολεία και σας υπενθυμίζω ότι όταν γίνεται λόγος για ασφάλεια Μιλούμε για την ασφάλεια των πληροφοριών, γιατί υπάρχουν κύβερνο επιθέσεις και σημαντικών πληροφοριών. Ασφάλεια ε, του υλικού πληροφορικής γιατί είναι συστηματικές οι επιθέσεις που απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μιλούμε επίσης για την ασφάλεια των προσώπων και κτηρίων. Προτείνω να εγκρίνουμε το συντομότερο δυνατό και το γρηγορότερο δυνατό το περιεχόμενο του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού ε, υπαριθμών 3 του 2016 για την ασφάλεια των θεσμικών οργάνων. Είναι επίγον και συμφωνώ με την πρόταση του συναδέλφου Ζεγάρ Ντεπρέ. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, επομένως θετική η γνωμοδότηση για το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθμών 3 που ε, ενισχύει την ασφάλεια των οργάνων. Ο κύριος Ντεπρέ, παρακαλώ. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, αλλά είμαι συνεισηγητής. Γιατί η πρότασή μου για την πρόταση της Επιτροπής επηρεάζει, είναι μια πρόταση αυτή της Επιτροπής που επηρεάζει τον εαυτό της, αλλά και τον προπολογισμό των άλλων θεσμικών οργάνων, όπως και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα προτιμούσα να έχουμε συζήτηση και κλεισμένα το θυρών, κύριε Πρόεδρε, γιατί υπάρχουν κάποια ζητήματα που είναι αρκετά λεπτά κατά την άποψή μου. Θα έχουμε συζήτηση και κλεισμένα το θυρών, λέει ο Πρόεδρος, στο τέλος της συνεδρίασης το απόγευμα. Μπορούμε να περιμένουμε. Καλώς. Ε, χωρίς να προδικάσω λοιπόν ε, τι θα πει ο κύριος Ντεπχέ στη συνεδρίαση και κλεισμένων των θερών. Εάν κανείς άλλος δεν ζητά το λόγο, θεωρώ ότι η Επιτροπή μας μπορεί να στηρίξει τη θέση του Γενικού Εισηγητή. Για τους προσανατολισμούς, λέω, του Ζωζέ Μανουέλ, για τις γενικές γραμμές. Ε, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Ο κύριος Ντεπρέ. Ναι, αλλά η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διορθώνει τον προϋπολογισμό της ΙΔΙΑΣ αλλά και τον προϋπολογισμό άλλων θεσμικών οργάνων δεν είναι μια πρόταση ε, διαιρετέα. Ε, πρέπει συνολικά να αποφανθούμε και να συζητήσουμε. Εν πάση θα επανέλθουμε, λέει ο Πρόεδρος. Καλώς. Ζωζέ Μανουέλ Φερνάντε, είστε εισηγητή και για τις εξελίξεις και τις ενδυνάμει τροποποιήσεις και προσαρμογές της ε, θεσμικής, υφιστάμενης θεσμικής δομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα το πρωί με τη συζήτηση που είχαμε ε, Είδαμε ότι έχει έρθει πλέον η στιγμή, είναι κατάλληλη στιγμή για να εξελιχθούν τα θεσμικά όργανα για να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της Ευρώπης και των Ευρωπαίων πολιτών. Σωσέ Μανουέλ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης η διαπίστωση είναι απλή. Για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει τις δικές της προκλήσεις, τις οποίες καλείται να, ε, ε, τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει, δηλαδή να πετύχει για παράδειγμα τους στόχους της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020, για να ανταποκριθούμε λοιπόν στις προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών, δεν μπορούμε να έχουμε προπολογισμό που να είναι 1% του ακαθάριστου εγχώριου εισοδήματος. Έχουμε στόχους φιλόδοξους αλλά και μεσοπρόθεσμους. Αμφότεροι είναι φιλόδοξοι ούτως ή άλλως και οι μακροπρόθεσμοι και οι μεσοπρόθεσμοι. Είναι αδύνατο να επιτευχθούν με τέτοιο προϋπολογισμό. Και σε ό,τι αφορά τα θέματα του προϋπολογισμού, πράγματι πρέπει να φτάσουμε σε ένα αληθινό σύστημα ίδιων πόρων, πραγματικό σύστημα ίδιων πόρων, με απλότητα, με διαφάνεια, με ισονομία, με ισότιμη αντιμετώπιση, ένα σύστημα ευανάγνωστο, εύληπτο από τους Ευρωπαίους πολίτες. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, θα πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε ε, περικοπές, αντισταθμίσεις, αποζημιώσεις, που το μόνο που κάνουν είναι να περιπλέκουν το σύστημα και να μειώνουν τη διαφάνειά του. Και να μειώνουν και την ισότιμη αντιμετώπιση. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει όσο δυνατόν περισσότερη ευελιξία και να μην ξεχνούμε τα ποσά που έχουν καθοριστεί, γιατί δεν έχει νόημα να προσδιορίζουμε συγκεκριμένες αναλήψεις υποχρεώσεων και στη συνέχεια να ε, τις αλλάζουμε και να απελευθερώνονται κονδύλια. Γιατί έτσι έχουμε θεσμεύσεις, commitments που χάνονται. Γιατί είναι κονδύλια τα οποία ε, όταν δεν κινητοποιούνται ως ε, υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών ουσιαστικά χάνονται και τελικά υπάρχει πλεόνασμα στον προπολογισμό και όλα αυτά επιστρέφουν στα κράτη-μέλη ως έσοδα. Ενώ είναι έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να παραμείνουν για αυτήν και για το δικό της προϋπολογισμό. Θα πρέπει να τηρείται η αρχή της ενότητας του προϋπολογισμού. Η ενότητα δεν θα πρέπει τελικά να μεταφράσετε σε μείωση του προπολογισμού γιατί υπάρχουν κονδύλια που δεν χρησιμοποιούνται και επιστρέφονται στα κράτη-μέλη. Έχουμε χρηματοδοτικά εργαλεία ε, κατά πιστεύματα διαφόρων ειδών μέσα που έχουμε δημιουργήσει κυρίως για να αντιμετωπίσουμε την προσφυγική κρίση αλλά και, άλλα, και άλλες προτεραιότητες. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει όλοι αυτοί οι οικονομικοί ε, και χρηματοδοτικοί μηχανισμοί να υπάρχουν στο προπολογισμό για να ασκηθεί ο κατάλληλος κοινοβουλευτικός έλεγχος και να νομοποιηθεί ο προπολογισμό. Περιμένω λοιπόν τη συνεισφορά των συναδέλφων για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης και πιστεύω ότι οι τροπολογίες ε, αν δεν απατώμε, μπορούν να κατατεθούν μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Περιμένω λοιπόν τη συνεισφορά σας υπό τη μορφή τροπολογιών και θα προσπαθήσω να συμπεριλάβω όσο περισσότερες μπορώ. χωρίς να ξεπεράσω ε, το μέγεθος ε, του κειμένου που μου επιβάλλεται. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος. Και εγώ έχω κάτι να αλλάξω. Δεν είναι 8 Σεπτεμβρίου, είναι 5 Σεπτεμβρίου η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών, λέει ο πρόεδρος. Στις 5 Σεπτεμβρίου. Εκτός μικροφώνου ο κύριος Φενάντες. 5 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα ε, είναι η καταληκτική προθεσμία. Ο κύριος Φερναντές στην ημερήσια διάταξη το αναγράφει ότι είναι μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου. Είναι τυπογραφικό λάθος στην ημερήσια διάταξη. 5 ε, Σεπτεμβρίου είναι τελικά η καταληκτική προθεσμία. Ευχαριστώ τον κύριο Φερναντές. Ποιος θέλει το λόγο. <clears throat> Κύριε Βιώτη, ευχαριστώ τον συνάδελφο Φερνάντες <clears throat> και για μένα λέει 5 <clears throat> Σεπτεμβρίου. Γιατί πρόκειται για συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν τον προπολογισμό και συμφωνώ ιδιαίτερα για το ότι γίνεται ανάφορα την ε, ε, επέκταση του προπολογισμού και θα πρέπει να το συζητήσουμε και με την ομάδα μου σε ό,τι αφορά το κατά πόσον συμφωνούμε την επιστροφή των ε, κονδυλίων στους εθνικούς προϋπολογισμούς και φυσικά και το κατά πόσον συμφωνούμε και με την αρχή της δίκαιης επιστροφής και θα δούμε λοιπόν όταν θα μας ανακοινώσετε και την ημερομηνία για την υποβολή των τροπολογιών σε ό,τι αφορά τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Τζάε. Έχω κάποια σχόλια τα οποία θα υποβάλω υπό μορφή τροπολογιών, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει πιο συγκεκριμένη παράγραφος για τα συνέπειε του Brexit. Ευχαριστώ. Θέλει κάποιος άλλο το λόγο. Κοιτάξτε, έχω ένα σχόλιο να κάνω. Ο προπολογισμό μας είναι κατά βάση ανα διανεμητικός. Οι στόχοι που επιδιώκει το θεσμικό έργο, ε, όργανο ε, εφαρμόζονται και επιτυχάνονται με την εφαρμογή του προϋπολογισμού. Και πρέπει ο προϋπολογισμός λοιπόν να ε, περιλαμβάνει τα μέσα που θα επιτρέψουν στο θεσμικό όργανο να πετύχει τους στόχους του και είναι θέμα ε, κυριαρχίας που μοιραζόμαστε. Και αυτό ισχύει στο νομισματικό επίπεδο. 5 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα. Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή στις 26 ή στις 29 Σεπτεμβρίου. Ο κύριος Τάραντ είναι μαζί μας να μας παρουσιάσει την έκθεσή του. για την εταιρική σχέση, τη σύμπραξη για τη βιώσιμη αλληλεία. Όχι, αλλιώς τότε θα εξετάσουμε αργότερα αυτό το φάκελο. Έτσι κερδίζουμε ενδεχομένως λίγο χρόνο. Πάμε στην εφαρμογή του προγράμματος «Η Ευρώπη για τους πολίτες». Συνάδελφος Χριστοφόρου. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ανταποκριθώ στο έτοιμα σας και θα κερδίσουμε ακόμα περισσότερο χρόνο για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπήρξε κανένα προσχέδιο ούτε έκθεση ούτε αναφορά από καμιά επιτροπή ούτε από την Επιτροπή Πολιτισμού και εκ των πραγμάτων μου ήταν αδύνατο να συντάξω οποιαδήποτε γνωμοδότηση. Το ευχάριστο είναι ότι η κατάθεση τροπολογιών είναι μετά από 20-21 μέρες, 21 Σεπτεμβρίου και θα καλέσω τους συναδέλφους να με υποβοηθήσουν σε αυτό το έργο με τις τροπολογίες και ό,τι άλλο θα ήθελαν να καταθέσουν για να βελτιώσουμε το υπό ε, σύνταξη ε, σχέδιων τόσο σε επίπεδο έκθεση όσο και σε γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Euh, c'est un rapport, euh, une communication Ευχαριστώ πολύ. Ήσασταν πολύ συγκεκριμένο. και σας ευχαριστώ θερμά. Ποιος θέλει το λόγο? θα ήθελα ο προϋπολογισμός να είναι εύληπτος και κατανοητός για τους Ευρωπαίους πολίτες, για το θέμα της Ευρώπης, για τους πολίτες, για αυτό το πρόγραμμα και αυτή την έκθεση. Εάν δεν θέλει κανείς το λόγο για το σημείο 9, να σας πω ότι καταληκτική προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 18η Οκτωβρίου το μεσημέρι, στις 12 το μεσημέρι. 18 Οκτωβρίου μέχρι τις 12 το μεσημέρι έχουμε λοιπόν 6 εβδομάδες σχεδόν. Ε, μπορεί ο κύριος Εστέμπαν Κονζάλες να μας μιλήσει για την Ευρωπαϊκή Ένωση της Άμυνας. Το θέμα που αναφέρθηκε σήμερα το πρωί στα σχόλια του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2017 μιλήσαμε για μια προπαρασκευαστική ερευνητική δράση για την Ευρώπη της Άμυνας. Παρακαλώ κύριε Κονσάλε Σπόνζε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας παρουσιάσω την γνωμοδότηση που προτείνω σε αυτή την Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση της Άμυνας. Ε, το προσχέδιο έχει πέντε παραγράφους και προσπαθώ εκεί να συνοψίσω τα θέματα που μας αφορούν περισσότερο και να περιοριστώ στην οπτική γωνία του προϋπολογισμού. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συλλογιστεί το πώς θα φτάσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Άμυνας και πρέπει να είναι προτεραιότητά μας αυτή με στρατιωτικές δαπάνες 200 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, παρόλα αυτά ε, έχουμε κατακαιρματισμό του προϋπολογισμού, κατακαιρματισμό των δαπανών και άρα σπατάλες. Θα έχουμε τεράστια εξοικονόμηση. Αν έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση της Άμυνας, θα έχουμε καλύτερες επενδύσεις και καλύτερη έρευνα μπορούμε να εξοικονομήσουμε 26 δις από τα 200 ε, δις που σπαταλώνται αυτή τη στιγμή και να φτάσουμε και σε εξοικονόμηση 30 δις. Επομένως όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για να, και θα πρέπει να κινητοποιήσουμε διαφόρους μηχανισμούς όπως είναι η δομική μόνιμη συνεργασία της Συνθήκης Λισαβόνας και άλλα ε, θέματα. Στο προσχέδιο ζητώ να διευρυνθεί ο μηχανισμός Αθηνά και να μη χρηματοδοτεί τελικά το κάθε κράτος το δικό του στρατιωτικό προπολογισμό, αλλά να έχουμε κοινό. Έχουμε πολλά ερευνητικά προγράμματα, θα πρέπει να τα ενισχύσουμε, να μοιραστούμε πόρους και προτείνονται και διάφορες προτάσεις για το μέλλον. Δηλαδή σε αυτή τη γνωμοδότηση θεωρώ ότι έχει έρθει η στιγμή να ξεπαγώσει ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Άμυνα για να λυθεί και το πρόβλημα της ελλειπούς επένδυσης στις αμυντικές ικανότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα πρέπει να έχουμε ευρωπαϊκό εξάμεινο για την άμυνα, όπως έχουμε για τις οικονομίες, και έτσι τα κράτη-μέλη να συντονίσουν τις διαδικασίες τους μέσω μιας ανοιχτής διαδικασίας, στην οποία να παρεμβαίνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και παραμένω στη διάθεσή σας για σχόλια, για προτάσεις. Σίγουρα μπορεί να βελτιωθεί αυτό το προσχέδιο και να αντικατοπτρίσει ε, τις θέσεις όσο να το περισσότερο. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος και εγώ ευχαριστώ τον κύριο εισήγητη. Ένα σχόλιο, Πρόεδρε, το οποίο είναι γενικού χαρακτήρα θα έλεγα για τα θέματα του προϋπολογισμού. Σήμερα το πρωί είδαμε όταν συζητούσαμε για τον προϋπολογισμό του 17 ότι το θέμα αυτό είναι κάτι το οποίο απασχολεί συνεχώς τη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο <clears throat> και με αυτή την προπαρασκευαστική δράση η οποία είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες της Ένωσης στο μέλλον. Χωρίς να μπω τώρα στην ουσία, για μια ακόμη φορά έχουμε μια νέα προτεραιότητα <clears throat> και θα πρέπει να υπάρξει μια νέα μορφή χρηματοδότησης. Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα τα οποία να αντιστοιχούν με τις προτεραιότητες που αποφασίζονται. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να υπογραμμίσουμε το θέμα της χρηματοδότησης αυτής της νέας προτεραιότητας που θα βρούμε τα χρήματα και ελπίζουμε τα κράτη-μέλη να επιδείξουν την ευθύνη που απαιτείται για να βρουν τα χρήματα αυτά. Τώρα γιατί από κοινή προσπάθεια, η κοινή προσπάθεια πράγματι και θα βελτιώσει τις δυνατότητες μας και θα κοστίσει λιγότερο. <clears throat> θα πρέπει να περιμένουμε λοιπόν τις απόψεις Συμβουλίου. Έτσι ώστε να μην υπάρξουν περικοπές και να βελτιώσουμε λοιπόν τους πόρους και να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα χρήματα των φορολογουμένων. Ευχαριστώ. Ο εισηγητής. Συμφωνώ με την άποψη της κυρίας Γουαδιασάβαλ και θα ήθελα η άποψη αυτή να περιλαμβάνεται καλύτερα στην νομοδότησή μου για να τη βελτιώσει ακόμα περισσότερο. Το θέμα είναι να δούμε ποιε είναι τα θέματα κυριαρχίας τα οποία θα ασκηθούν πιο αποτελεσματικά εφόσον αναλυθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο από ό,τι σε εθνικό. Το θέμα της άμυνας είναι σημαντικό θέμα, το ίδιο και η διπλωματία. <clears throat> Θα πρέπει να δούμε ας πούμε τι κτίρια διπλωματικά υπάρχουν από τις χώρες στον κόσμο και καταλαβαίνετε ότι το θέμα της αμοιβεοποίησης των χώρων των διπλωματικών υπηρεσιών θα προσφέρει οικονομίες πολλές εξοικονομήσεις πολλές, συγγνώμη, στα κράτη-μέλη και στην ίδια την Ένωση. Και εδώ μπορούμε να κινητοποιήσουμε και την κοινή γνώμη, γιατί οι πολίτες το καταλαβαίνουν αυτό. Αν υπήρχε μια ξεκάθαρη θέση για το Ιράκ, ας πούμε, για τη Λιβύη, για τη Συρία, ίσως να μην γνωρίζαμε σε τέτοιο βαθμό μεταναστευτικές ροές. Εγώ πρόσφατα είχα πάει στην Μέση Ανατολή και πρέπει να πούμε ότι οι απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το όραμα της Ευρώπης δεν είναι ξεκάθαρες. Και οι εκπρόσωποι μας εκεί κάνουν ό,τι μπορούν με μια σχετική αποτελεσματικότητα κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Λοιπόν δεν ξέρω αν θέλει κάποιος άλλος το λόγο για την έκθεση González Pons. <coughs> Διευκρινίζω ότι η προθεσμία είναι η 8η Σεπτεμβρίου, σε μια εβδομάδα. Και θα υιοθετήσουμε το σχέδιο αυτό στις 10 ή στις 11 Οκτωβρίου στη συνεδρίασή μας. Επέστρεψε ο κύριος Τάραντ. Έχει το λόγο. για τις απόψεις του για την αλλιευτική συμφωνία με τα νήσους Κουκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που ε, καθυστέρησα, δεν ήμουν εδώ όταν αναφερθήκατε την πρώτη φορά στο ζήτημα αυτό. Έχουμε προεδρικές εκλογές στην Εσθονία και με κάλεσαν στο τηλέφωνο γιατί ζητούν την εμπειρογνωμοσύνη μου. Εν τω μεταξύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δουλέψει πολύ σκληρά για να διασφαλίσει τα αλλιευτικά δικαιώματα των Ευρωπαίων αλλιέων στις εξόχως απόκεντρες θάλασσες και στα νησιά Κουκ και έχουμε μία συμφωνία με τις νήσους Κουκ και αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληρώσει 2,87 εκατομμύρια σε βάθος 8 ετών και θα έχουμε ένα κόστος για τον προϋπολογισμό 350.000 ευρώ ετησίως και μπορούμε να αλλιεύουμε 7.000 ε, τόνους ετησίως. Ένα κιλό ψαριού μας στοιχίζει 5 ευρώ. Ζητώ από όλους να το εγκρίνουν. Και θα ψηφίσω κατά μόνο αν τα εστιατόρια στις Βρυξέλλες ε, αυξήσουν τις τιμές των ψαριών. Εν πάση περιπτώσει 5 ευρώ ε, το κιλό του ψαριού θα αγοράζουμε. Είναι η τιμή που πληρώνουμε για να μπορούμε να αλλιεύουμε εκεί. Ο καταναλωτής αναλαμβάνει το κόστος του ε, ψαριού που πληρώνει ο, ο καταναλωτής, ο φορολογούμενος το αναλαμβάνει. Λοιπόν, καταληκτική προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Το μεσημέρι στις 12, 7 Σεπτεμβρίου. 10 ή 12 Οκτωβρίου θα ψηφίσουμε. Η Επιτροπή Αλίας θα ασχοληθεί με το φάκελο και θα το εγκρίνει στις 9 ή στις 10 Νοεμβρίου και στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου θα εγκριθεί ε, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο σύσσωμο θα έχει την ευκαιρία να αποφανθεί επί ε, του κειμένου αυτού. Και αντίθετα με ό,τι είπα, δεν αντιστρέψαμε, δεν εξετάσαμε το 12 πριν από το 11. Ο κύριος Βιώτη έχει το λόγο για την επένδυση στην ανάπτυξη, στην οικονομική μεγέθυνση, στην απασχόληση. Θα είμαι σύντομος. Είναι γνωμοδότηση για την έκθεση της Επιτροπής Ρέτζη στα πλαίσια του νέου κανονισμού των διαφορετικών ταμείων και με βάση τη μελέτη η οποία παρουσιάστηκε και εφαρμόστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεση αυτή συγκεντρώνουμε την προσοχή μας πάνω στα δημοσιονομικά θέματα. Τρία είναι αυτά. Το θέμα του υπολογισμού των επιδόσεων της εφαρμογής των ταμείων, οι χρηματοδοτήσεις σε σχέση με τις ευρωπαϊκές παρεμβάσεις και η προσθετικότητα ανάμεσα στα διαφορετικά ταμεία και το στρατηγικό ταμείο επενδύσεων. Πάνω σε αυτό έχει μιλήσει ο Επιτροπός κατά είναι επανειλημμένα, έχει ενδιαφέρον. Τέλος, ζητάμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει συγκεκριμένες πληροφορίες το ταχύτερο δυνατόν για τις χρηματοδοτικές συνέπειες του Brexit και τη νέα Ευρώπη των 27. Η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι η 8η Σεπτεμβρίου 12η Μεσημβρινή. Ευχαριστώ κύριε Βιώτη. Θα ήθελε κάποιος άλλος το λόγο <clears throat> για την έκθεση του κυρίου Βιώτη, ο κύριος Όλμπριχτς. Εξ ονόματος του ΕΤΚ να πω ότι η έκθεση αυτή αποτυπώνει και τα όσα συζητήσαμε στην αρχή της συζήτησης για τον προπολογισμό σε ό,τι αφορά τα, τους πόρους για το ΕΕΣΥ, για το μέλλον και πώς θα ασφαλιστούν αυτοί. Πρόκειται για ένα θέμα, ένα πρόβλημα ε, συμπληρωματικότητα σε ό,τι αφορά τα ταμεία αυτά. Ιδιαίτερα κοιτώντα ε, τι ανησυχίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την πρόταση για την παράταση του ΕΦΣΥ, Θα πρέπει να είναι σαφέ, λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά τα θέματα συμπληρωματικότητας δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Υπάρχουν προτάσεις, αλλά δεν υπάρχει σαφής πρόταση για συγκεκριμένους ρόλους. Ένα λοιπόν στοιχείο είναι το θέμα της ε, σχέσης ε, μεταξύ εύση και των άλλων ε, ταμείων και να τονίσω και αυτά που είπε ο συντονιστής ο κ. Φανής στην ερώτηση σε ό,τι αφορά την αποδοτικότητα και την απόδοση του ΕΦΣΙ Ενδεχομένως, να πρέπει να προτείνουμε μια διαφορετική διατύπωση σε ό,τι αφορά τη σχέση της απόδοσης των ε, ταμείων ΕΦΣΙ και το θέμα ε, του θέματος της αξιολόγησης. Θα δούμε λοιπόν πώς θα δημορφωθεί αυτό στο μέλλον. Ενδεχομένως λοιπόν να χρειαστεί μια διαφορετική διατύπωση για την ε, έκθεση και ήθελα απλά να ζητήσω συγγνώμη για την απουσία του συντονιστή μας. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Θα τα συζητήσουμε αυτά και στην κοινή ε, συνάντηση. Αν δεν επιθυμεί κανεί άλλο το λόγο για τα θέματα αυτά. Η κυρία Χόλμαϊρ, πού βρίσκεται. Μόλις έρθει θα τη δώσουμε κατευθείαν το λόγο. Για ένα θέμα το οποίο το έχουμε εξετάσει σε διάφορες περιστάσει και στήχησε στο σε πόντους. Μητρό, εισόδου, εξόδου. Je salue Madame Holmeyer. Je l'invite à s'installer. Καλώς ορίσατε κύριε Holmeyer, καθίστε. Βλέπω ότι οι διακοπές σας ήταν πολύ καλές, Αυτή την εντύπωση έχω. Ίσως σύντομες. Έχετε το λόγο κυρία Χολμάγερ, παρακαλώ. Πολύ σας ευχαριστώ πρόεδρε. Είσοδος, έξοδος, σύστημα εισόδου-έξοδου. Γνωμοδότηση προς την ε, αρμόδια Επιτροπή, ε, Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Το σύστημα λοιπόν εισόδου-εξόδου. Αυτό που εμάς μας απασχολεί ω Επιτροπή Προπολογισμού είναι τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε και στο σύστημα ΣΥΣ, για παράδειγμα. Το κόστος έχει αυξηθεί εκθετικά. Τότε λοιπόν είχαμε αποφασίσει επί ενός συστήματο, χωρί να ξέρουμε απαραίτητα τι μπορούσαμε να περιμένουμε από το σύστημα αυτό και χωρί να έχουμε και ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. χωρίς να έχουμε συμφωνήσει κάτι συγκεκριμένο με τα κράτη-μέλη τότε. Και αυτό λοιπόν σήμερα ότι δεκαπλασιάστηκε το κόστος. Αυτό ασφαλώς ε, προκάλεσε και μεγάλο θυμό, οργή, προβλήματα τεχνικά, τεχνικά με τα κρατημέλη, αντιπαραθέσεις μεταξύ των κρατών μελών, αντιπαραθέσεις στο στερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί μπλέχτηκαν και δύο διαφορετικές γενετικές διευθύνσεις, οι οποίες δεν ε, συμφωνούσαν απαραίτητα και όλα αυτά λοιπόν οδήγησαν σε σημαντικά προβλήματα. Και ως εκ τούτου πιστεύω από πλευρά τη Επιτροπή μα, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο εξή. Αν είναι να εισαχθεί ένα τέτοιο σύστημα, θα πρέπει να εισαχθεί με πολύ στοχοθετημένο τρόπο. Θα πρέπει να διευκρινιστούν τεχνικέ λεπτομέρειε και θα πρέπει να συμφωνηθούν αυτά με τα κρατημέλη που ήδη έχουν τέτοια συστήματα, γιατί υπάρχουν κρατημέλη που έχουν τέτοια συστήματα. Θα πρέπει να ξέρουμε λοιπόν τι υπάρχει τι διατίθεται από τεχνική άποψη, ποιε είναι οι επαφέ, ποια είναι τα περιεχόμενα. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να είναι τεχνικός πόσο συμβατά προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κοινό σύστημα. Και θα πρέπει να σκεφτούμε στη συνέχεια το τι γίνεται με τα κρατημέλη που δεν έχουν ακόμα τέτοιο σύστημα. Τι προποθέσει θα πρέπει να πληρούνται για να δημιουργηθούν αντίστοιχα συστήματα στα κρατημέλη αυτά και το πώ τα 28 αυτά συστήματα θα μπορέσουν να εναρμονιστούν με κάποιο τρόπο. Μου κάνει εντύπωση ότι δεν προβλέπεται κανένας μηχανισμός ε, για το τι θα συμβεί αν κάποιο κράτος μέλος δεν έχει χρηματοδότηση, δεν έχει προσωπικό, δεν έχει εμπειρογνώμονες. Θα μείνουμε όλοι πίσω λόγω ενός κράτους μέλους που δεν τα εφαρμόζει αυτά και θα καθυστερεί τους 27 άλλους. Εδώ λοιπόν δεν προβλέπεται κανένα σύστημα. Τι θα γίνει λοιπόν αν ένα κράτος μέλος τυχόν δεν τα βγάλει πέρα για το χύψη λόγο. Για παράδειγμα, επειδή η Ελλάδα ενδεχομένω μπορεί να πει ότι δεν το αντέχουμε αυτό τώρα οικονομικά στην παρούσα φάση και δεν το σηκώνουμε. Τι θα γίνει και τι θα γίνει και με την αρχή που τούτη δεν δημιουργούμε επιπλέον χρέη κτλ. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώ θα προβλεφθεί αυτό ο μηχανισμό προκειμένου να έχει και νόημα από οικονομική και δημοσιονομική άποψη. Θα πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε ε, τον δεκαπλασιασμό του κόστους. Αυτά θα πρέπει να τα ξέρουμε πρωτού προκηρυχθούν τα έργα αυτά. Για να μην ε, βρεθούμε σε δυσχερή κατάσταση υπό πλευρά ε, δημοσιονομική και να έχουμε προβλέψει το ΑΒΓΔ και να έχουμε χάσει όλο το υπόλοιπο αλφάβητο. και θα πρέπει να θα συζητήσουμε αυτά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί υπάρχει μια πολύ γενική, ένα πολύ γενικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά το κόστος. Δεν ξέρουμε συγκεκριμένα τι θα επιβαρύνει τα κρατημέλη, ε, πόσο θα επιβαρύνει, τι θα επιβαρύνει τον προπολογισμό. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε επακριβή στοιχεία στη διάθεσή μας και για την δημοσιονομική πτυχή ε, μεσοπρόθεσμα για τη δημιουργία των συστημάτων, αλλά και μακροπρόθεσμα για τη διατήρηση, τη συντήρηση του συστήματος, την ανανέωση του συστήματος όταν θα έλθει ο, η χρονική στιγμή. Χρειάζεται λοιπόν ε, ένα τέτοιο πίνακα. Και στο ΣΥΣ παρουσιάστηκα, όπω σα είπα, ότι έχει προβλήματα, γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει μεγαλύτερη τεχνική ανάλυση για το ποιε θα είναι οι συνέπειε στον προπολογισμό. Αυτά θα ήταν τα πιο σημαντικά σημεία σε ό,τι αφορά τις δημοσιονομικές επιπτώσεις ενός τέτοιου συστήματος. Ευχαριστώ, κυρία εισηγήτρια. Ο κύριος Ντεφρέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ήμουν παρόν όταν συζητήσαμε το σύστημα εισόδου-εξόδου και συμφωνώ πολύ με τη συνάδελφο κυρία Χολμάιερ. Έχω κάτι άλλο όμως να ρωτήσω. Το σύστημα που θα εφαρμόσουμε είναι ένα σύστημα που θα μας επιτρέπει να αναγνωρίζουμε όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών που μπαίνουν στο χώρο Σέγγεν και που βγαίνουν από αυτόν. Καλώς. Ως τέτοιο λοιπόν δεν έχει κανένα ενδιαφέρον εκτός εάν αυτά τα δεδομένα διασυνδέονται με άλλες βάσεις δεδομένων. Επομένως, ερωτώ, ερωτώ την κυρία Χολμάγερ. Στο σχέδιο που εγκρίνουμε αυτή τη στιγμή καθορίζουμε τις ε, διασυνδέσεις και τις ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων συστημάτων, το σύστημα πληροφοριών Schengen, την τράπεζα δεδομένων του Eurodac. Αν απλά καταχωρίζουμε ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει και δεν το συνδέουμε με τίποτα, είναι ανόητο είναι τεράστιο κόστος για να έχουμε καταλόγους ονομάτων χωρίς ε, να γνωρίζουμε κάτι για αυτούς. Μπορεί ίσως η Επιτροπή να απαντήσει. Και αν ε, είναι ναι η απάντηση, ε, με ποιο σκοπό και ποιου είδους δεδομένα θα διασυνδέονται με άλλες βάσεις και τράπεζες δεδομένων. Και αν δεν μπορεί η κυρία Χολμάγερ να απαντήσει, απευθύνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι προβλέπετε. Μπορεί να απαντήσει η κυρία Χολμάγερ. Πριν της δώσω όμως το λόγο, θα δώσω το λόγο στην κυρία Ταπαρντέλ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, εκ μέρους των σοσιαλιστών χαίρομαι διότι γίνεται αυτή η συζήτηση σήμερα και μπορούμε να έχουμε την αναθεώρηση του κανονισμού του 2013 για το σύστημα εισόδου και εξόδου όσον αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών που ε, διασχίζουν τα εξωτερικά σύνορα της ζώνης Σέγγεν. Θεωρούμε ότι αυτό το σύστημα είναι απολύτως απαραίτητο, αυτό ισχύει εδώ και καιρό και απαντά στα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή, η οποία χρειάζεται έξυπνα, ενιαία, ολοκληρωμένα σύνορα για να διαχειριστεί τη ροή των επισκεπτών, ε, τουριστών, αλλά και όλων όσοι διασχίζουν τα σύνορα ε, με ένα ρυθμό ε, συνεχή οι μεταναστευτικές αρχές μας λένε ότι τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους είναι στοιχειώδη. Πήγαμε στη Λαμπεντούζα πέρσι και είδαμε πόσο περιορισμένοι είναι οι πόροι και οι δυνατότητες. Οι διαδικασίες στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μία αποτελεσματικές και τα λάθη συσσωρεύονται. Και επιτρέψτε μου να κάνω μια παρένθεση σε σχέση με την τωρινή μας συζήτηση και να μιλήσω για το κεκτημένο Σέγγεν. Είναι ευκταίο να απλοποιηθεί το κεκτημένο Σέγγεν και η Ρουμανία και η Βουλγαρία πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να μπουν στο Σέγγεν. Θα πρέπει το Σέγγεν να είναι ισχυρό ο χώρος αυτός και να προσχωρήσουν σε αυτό όλες οι χώρες μέλη. Έχουν αλλάξει διάφορα πράγματα στο υφιστάμενο πλαίσιο, στην υφιστάμενη χρονική συγκυρία και σε θέματα ασφαλείας. Η καλή διαχείριση των συνόρων είναι απαραίτητη για την εσωτερική ασφάλεια και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Θα πρέπει να έχουμε ένα κεντρικό, ενιαίο και απλουστευμένο σύστημα για την ανταλλαγή των πληροφοριών και των δεδομένων. Και τέλος, θα πρέπει να εφαρμόσουμε και να προβλέψουμε να υπάρξουν οι απαραίτητες δράσεις για να εγγυηθούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα των επισκεπτών, των περιηγητών, των ταξιδιωτών, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ειδικότερα σήμερα με το σημερινό εφιστάμενο πλαίσιο η, λύση πρέπει να είναι ευρωπαϊκή και όχι κόψε ράψε ένα μοσαϊκό από τις εκατατόπους λύσεις των διαφόρων κρατών μελών. Θα πρέπει να νιώθουν, σε... να νιώθουν ασφάλεια οι επισκέπτες και να μην είναι η Ευρώπη ένα κλειστό φρούριο στον οποίο να μην μπορεί να έχει πρόσβαση κανείς. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος, ποιος άλλος θέλει το λόγο παρακαλώ. Θα ήθελα και εγώ να απευθύνω ένα ερώτημα στην κυρία Χολμάγερ. Όλα τα κράτη-μέλη θα έχουν τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές για το αρχείο τους, για το μητρό τους, για να μην υπάρχουν δυσκολίες σύνδεσης μεταξύ των διαφόρων συστημάτων και αυτά θα συνδέονται με το Μητρό των Προσφύγων. Και προετοιμάζουμε έτσι την αναθεώρηση του Δουβλίνου, γιατί στη Σικελία πέρσι όταν πήγαμε είδαμε ε, πόσο μη αποτελεσματικό και μη λειτουργικό είναι το σύστημα του Δουβλίνου, η συμφωνία του Δουβλίνου. Είτε καταχωρίζει κανείς, είτε δεν τα χωρίζει, γιατί ορισμένοι μετανάστες δεν καταχωρίζονται γιατί δεν θέλουν να παραμείνουν στην Ιταλία όσο ωραία και είναι αυτή η χώρα. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Όλη αυτή η δομή είναι που τίθεται ένα αμφιβόλο. Και αν για την υποδοχή των προσφύγων έχουμε τόσες ερμηνείες του δικαιώματος ασύλου όσες χώρες μέλη έχουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε δεν λύνεται ποτέ κανένα πρόβλημα. Και νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες το καταλαβαίνουν αυτό, θα το καταλάβουν και θα ε, είναι στο πλευρό μας. Κλείνω την παρένθεση και δίνω τον λόγο στην κυρία Χολμάγια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, το ερώτημα του κατά πόσο υπάρχει υποχρέωση για την καταχώρηση των κρατών μελών. Ε, αυτό υπάρχει ήδη ως υποχρέωση. Η εφαρμογή είναι αυτή που διαφέρει. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, δεν επεξεργαστεί, δεν ε, εκτέλεσε δεν, αυτή την, ε, αυτό το καθήκον. Και στην Ιταλία υπήρχαν προβλήματα, αλλά και στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρχαν ε, πολλές ε, χώρες που δεν ήταν στα σύνορα, ήταν η Ουγγαρία, Αυστρία, Σλοβενία, η Γερμανία, διάφορες χώρες, η Γαλλία που δεν τήρησαν απόλυτα το Eurodac. Και αυτό για διάφορους λόγους ε, με διάφορες δικαιολογίε ότι δεν θέλουν να καταχωρίζονται οι μετανάστες, οι πρόσφυγες ε, και έχω την εντύπωση ότι δεν υπήρξε μια νέα στρατηγική, αλλά η θέληση, η προθυμία από πλευρά των κρατών μελών να γίνει η καταχώρηση έχει αυξηθεί. Γιατί είναι τεράστια η κίνδυνη τη ε, μετακίνηση των ατόμων. Και υπάρχουν και στοιχεία ότι που καταδεικνύουν ότι αυτοί οι άνθρωποι σε πολλές περιπτώσεις εκλειστρούν στην εγκληματικότητα από την οποία και δεν βγαίνουν σε πολλές περιπτώσεις το οργανωμένο έγκλημα, Πολύ νέοι ιδιαίτερα, είτε είναι καταναγκαστική πορνεία, είτε είναι άλλοι ε, τομείς ε, αυτοί, αλλά Στη συνέχεια ο κόσμος ε, πώς θα πάει στην αστυνομία και θα στραφεί στην αστυνομία όταν φοβάται ότι ε, θα τον αναγνωρίσουν και ότι είναι δεν έχει καταχωριστεί και δεν έχει μπει σε κανένα σύστημα και είναι λίγο φαύλο κύκλο αυτό. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να το σπάσουμε αυτό το φαύλο κύκλο. Αυτή η έλλειψη καταχώρηση δεν είναι κάτι φιλικό προ τον άνθρωπο, όχι, είναι επικίνδυνο αυτό για τον κόσμο, γιατί δεν είναι... Είναι ανώνυμοι, δεν έχουν σε ποιον να στραφούν, δεν έχουν σε ποιον να αποτανθούν και αυτό συνεπάγεται τεράστιους κινδύνους. Και αυτό σε κάποιες περιπτώσεις νομίζω ότι παρανοείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ε, φιλελευθερισμός. Το λέω αυτό ξεκάθαρα. Λοιπόν, αυτέ οι υποχρεώσει θα πρέπει να ισχύουν για όλα τα κράτη-μέλη. Και γι' αυτό λοιπόν στο σχέδιο γνωμοδότηση ε, ε, το υπογράμμισα αυτό, ότι όντω και στα 28 κράτη-μέλη θα πρέπει να εφαρμοστούν αυτά εγκαίρω. Εγκαίρω. Και θα απαιτήσουμε ένα τέτοιο μηχανισμό. Θα πρέπει λοιπόν και οι 28 να εφαρμόζουν το σύστημα αυτό και δεν έχει νόημα αν είναι... Αν υπάρχουν 3, 4, 5 που δεν εφαρμόζουν το σύστημα, δεν έχει νόημα οι υπόλοιποι 23 να κάνουν τέτοια καταχώρηση. Αυτό το σύστημα λοιπόν θα πρέπει να εφαρμοστεί είτε από όλους παράλληλα ταυτόχρονα, είτε να μην εφαρμοστεί καθόλου. Αυτό το μάθαμε και από τη Γυροντάκη, γιατί αυτό που είπε ο κ. Ζεραντεπρέ ήταν πάρα πολύ εύστοχο. Και σε ό,τι αφορά την διαλειτουργικότητα θα πρέπει να σας πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να υπάρχει διαλειτουργικότητα, αλλά υπάρχει και μία παρανόηση σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων. Προστασία των δεδομένων δεν σημαίνει ότι εκφράζουμε μια γενική υποψία κατά όλων που περνούν τα σύνορα, γιατί κοιτάμε για παράδειγμα κατά πόσον έχουν καταχωριστεί στο ΣΥΣ ή κάπου αλλού. Για παράδειγμα, αν ελέγχουμε αν υπάρχουν τα δακτυλικά αποτυπώματα α, ε, κάποιου ατόμου σε κάποια βάση δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή ενδεχομένω ε, να μην το επιτραπεί η είσοδο. Δεν πρόκειται λοιπόν για μια γενική υποψία. Ή θα πρέπει να σταματήσουμε και του φορολογικού ελέγχου. Δηλαδή, τι κάθε φορά που γίνεται φορολογικό έλεγχο, χωρί να υπάρχει συγκεκριμένα υποψία, τι σημαίνει ότι υποπτευόμαστε ε, όλους τους φορολογούμενους. Δεν θα κάνουμε δηλαδή και ελέγχους ε, ε, αλκοόλ και πνεύματος γιατί έτσι δεν θα κατηγορούμε όλους τους οδηγούς. Δηλαδή τι θα ελέγχουμε μόνο όσους ξέρουμε ότι έχουν πιει. Τι λογική είναι αυτή. Αυτό δεν μπορεί να ενταχθεί σε, μια, σε ένα πλαίσιο ελέγχου. Και ασφάλειας. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα σύστημα για να σταματάμε τους ε, δράστες ε, εγκληματικών ενεργειών στα σύνορα. Θα πρέπει να υπάρχει ένα καλό τεχνικό σύστημα το οποίο γρήγορα να επιτρέπει την αναγνώριση χωρίς να υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις. Αυτός είναι ο σκοπός του συστήματος. Αυτό θα πρέπει να εγγυηθούμε και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι σκοπεύει να κάνει για την διαλειτουργικότητα των βάσεων δεδομένων προκειμένου να επιτευχθούν αυτά όλα εγκαίρως. Και συμφωνώ λοιπόν απόλυτα με τον συνάδελφο Ντεπρέ. Για του συναδέλφους από του σοσιαλιστές και δε, δημοκράτες, το σύστημα εισόδου και εξόδου δεν συνδέεται απαραίτητα με το σύστημα Schengen σε ό,τι αφορά και τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Εδώ όμως τοποθετήθηκε με σαφήνεια το Κοινοβούλιο. Αν πληρώνουν τα κριτήρια, ευχαρίστω να μπει και η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Αυτό είναι θέμα μεταξύ των κριτών μελών, το οποίο δυστυχώ εδώ δεν μπορούμε να το ρυθμίσουμε με τις δικές μας ε, Όλα τα κράτη-μέλη, είτε είναι μέλη του Σέγγεν είτε όχι, θα πρέπει να θα συμμετέχουν στο σύστημα αυτό και αυτό δεν θα έπρεπε να ισχύει μόνο σύστημα για τις χώρες μόνο του Σέγγεν. Για όλες τις χώρες θα πρέπει να ισχύει. Μόνο τότε θα έχει αποτέλεσμα και νόημα ένα τέτοιο σύστημα. Συμφωνώ απόλυτα λοιπόν μαζί σας. Θα δώσω το λόγο τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αναφερθεί στο θέμα των ασυνόδευτων ανηλίκων. Υπάρχει εδώ ένα, πραγματικά μια παράνομη εμπορική δραστηριότητα. Κάποιοι λέγουν ότι είναι ανήλικοι, αλλά δεν είναι. Και οι συνέπειες είναι πάρα πολύ δύσκολες για τις, για τις δομές υποδοχής. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν να ξεκαθαρίσει λίγο αυτές τις απαράδεκτες μορφές σωματεμπορίας. Ο κύριος Φρέζα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. για το σύνολο λοιπόν των χωρών. Σας ευχαριστώ. Δεν έχω όλα τα στοιχεία για να δώσω λεπτομερείς απαντήσεις στον κύριο Ντεπρέ. Στόχος της διαλειτουργικότητας παραμένει ο στόχος. Θα στείλω γραπτός τις ε, λεπτομερείς συνθήκες οι οποίες ενδιαφέρουν και την Επιτροπή σας. Αφού όμως πάρω τα στοιχεία από τους συναδέλφους, δυστυχώς δεν τα έχω. Καλώς. <clears throat> Κύριε Χολμαϊέρ, θέλετε κάτι άλλο. <clears throat> Ακούσαμε τον κύριο Φρέζα μας είπε ότι δεν έχει τα απαιτούμενα στοιχεία για να δώσει απαντήσεις. Θα σας στείλει τις απαντήσεις αυτές και σε εσά και στον κύριο Ντεπρέ το ταχύτερο δυνατόν. Η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών προβλέπεται για τις 15 Σεπτεμβρίου, 12 το μεσημέρι, Α, κοιτάξτε, ίσως έκανα κάποιο λάθος. Ίσως έκανα κάποιο λάθος. Έγινε σήμερα μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Το σχέδιο εκθέσεως τέλος Σεπτεμβρίου, 26 ή 27. Και οι τροπολογίες θα κατατεθούν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άλλος που έχει ζητήσει το λόγο και γι' αυτό θα διακόψουμε τις εργασίες μας και θα ξεκινήσουμε σήμερα το απόγευμα στις 3.